Καλημέρα αγαπητοί κυρίες και ε, κύριοι συνάδελφοι. Ε, βρισκόμαστε πλέον στη δεύτερη μέρα της συνεδρίασης της Επιτροπής μας. Βλέπω πως ε, ακόμα συνεχίζονται πυρετοδός οι διαπραγματεύσεις εδώ στην αίθουσα. Έχουμε λοιπόν στην μερίσια διάταξή μας τον προϋπολογισμό του 2010 και τα ποσά τα οποία θα θέλαμε να δεσμεύσουμε για την Επιτροπή μας στον προϋπολογισμό του 2010. Για πολλούς είχαμε διακοπέ για το καλοκαίρι, αλλά κάποιοι από εμά συνέχισαν να εργάζονται. Ένας από αυτούς ήταν η Γιούτα Χάου και την ευχαριστούμε πολύ γιατί παρότι αναπληρωματικό μέλος έκανε όλη αυτή τη δουλειά για μας και θα της δώσουμε το λόγο ως ε, συντάκτρια, ώστε να μα ε, διευκρινίσει λίγο τα του προπολογισμού. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε και θα ζητήσω από όλους τους συναδέλφους εδώ να με επιτρέψουν να πω κάποια πράγματα παρότι δεν μιλούν όλοι τη γερμανική γλώσσα. Α, για να τα διευκρινίσω επειδή δεν με ξέρουν όλοι, να πω δύο-τρία πράγματα και να πω και δύο-τρία πράγματα για τον προπολογισμό γιατί ενδεχομένως κάποιοι συνάδελφοι να μην γνωρίζουν κάποια ζητήματα. Ε, κάποια βασικά ζητήματα. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες. Έχουμε 28 υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδρύματα, αρχές, για τα οποία είμαστε εμείς ως Κοινοβούλιο αρμόδιοι και κατά συνέπεια αναλαμβάνουμε είτε το συνολικό είτε τμήμα του προπολογισμού των υπηρεσιών αυτών. Η Επιτροπή ε, προβαίνει σε ένα προσχέδιο, στη σύνταξη ενός προσχεδίου του προϋπολογισμού και στη συνέχεια το Συμβούλιο, όπως πάντα, περικόπτει τον προϋπολογισμό, πράγμα που βέβαια πάντα ε, τρομοκρατεί λίγο ε, τους ε, εκπροσώπους των διαφόρων υπηρεσιών, αλλά δεν θα έπρεπε να το κάνει γιατί εμείς ε, επανερχόμαστε βέβαια πάντα στο προσχέδιο του αρχικού του προπολογισμού και με αυτό το πνεύμα θα πρέπει να γίνουν αντιληπτέ και δικέ μα προτάσει σε ό,τι αφορά του προπολογισμού των υπηρεσιών. Ταυτόχρονα υπάρχουν διαφορετικά είδη ε, υπηρεσιών, δηλαδή κάποιε ε, χρηματοδοτούνται, ε, ο προπολογισμό του χρηματοδοτείται και από τέλη τα οποία εισπράττουν κατά την άσκηση των εργασιών του. Για παράδειγμα, η υπηρεσία για τα χημικά προϊόντα στο Ελσίκη, η MEA, δηλαδή η αρμόδια υπηρεσία για τα φαρμακευτικά που εδρεύει στο Λονδίνο και αυτές οι υπηρεσίες είναι οι ε, ή μάλλον για αυτές τις υπηρεσίες δημιουργήθηκαν αυτά τα τέλη που σχετίζονται με το σκοπό τους. Δηλαδή, εάν δεν έχουν δαπανίσει το σύνολο του προϋπολογισμού τους σε ένα συγκεκριμένο έτος, δεν μπορούν να το καταθέσουν στην τράπεζα, αλλά μπορούν να ε, μεταβιβάσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το πλεόνασμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το διατηρεί ως απόθεμα και αν χρειαστεί η λόγω υπηρεσία τον επόμενο ε, χρόνο ε, ε, αυτό το ποσό, γιατί δεν επαρκεί ο προπολογισμό, μπορεί να το ζητήσει. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργεί προβλήματα η Επιτροπή. Έχει υπάρξει αυτό, δηλαδή και στην περίπτωση της EMEA ε, και στην ΕΕ είχε πάρει αυτό το ε, πλεόνασμα και το είχε συνυπολογίσει μέσα στο νέο προϋπολογισμό. Όχι όμως αυτά είναι επιπρόσθετα τέλη και ε, δεν μπορούμε βέβαια ποτέ εκ των προτέρων να ξέρουμε ποιο είναι το ύψος των τελών που θα εισπραχθούν μέσα σε ένα έτος και αυτό είναι μια καλή πρακτική, αποδεδειγμένη πρακτική. Ε, και γι' αυτό άλλωστε η ίδια πολιτική ακολουθείται και από τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό λοιπόν εγώ ουσιαστικά αυτό που κάνω είναι να προτείνω περισσότερα κονδύλια σε σχέση με αυτά που προτείνονται. Τώρα, ε, κάτι ακόμα για τι υπηρεσίε έχουν, υπάρχουν κάποια ε, ε, σχέδια σε ό,τι αφορά και το προσωπικό ε, στις υπηρεσίες. Εμείς προσπαθούσαμε εδώ και καιρό αγωνιστήκαμε μαζί με τις υπηρεσίες να ε, εκπονήσουμε σχέδια ανάπτυξη των υπηρεσιών τους ώστε να μπορέσουν και αυτές οι υπηρεσίες να λειτουργήσουν με αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό όμως σημαίνει ότι και εμείς ω Κοινοβούλιο δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε όπως θέλουμε μέσα σε αυτό το οργανόγραμμα των υπηρεσιών όχι, δεν μπορούμε εμείς να ε, θεωρούμε ότι γνωρίζουμε καλύτερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ακόμα και από το Διοικητικό Συμβούλιο ε, μιας υπηρεσίας πόσα άτομα χρειάζεται αυτή η υπηρεσία για να εκτελέσει σωστά τα καθήκοντά της. Άρα λοιπόν, οι τροπολογίες εκείνες οι οποίες αναφέρουν ότι θέλουμε δύο περισσότερες ε, θέσεις ε, εργασίας ε, για την υπηρεσία στο Ελσίνκι, δηλαδή για τα χημικά. Μία τέτοια τροπολογία δεν μπορούμε να τη δεχτούμε. Δεν έχει νόημα. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μία συγκεκριμένη τάξη με πειθαρχία σε ό,τι αφορά 28 διαφορετικές υπηρεσίες. Η κάθε υπηρεσία θα πρέπει, ξεκινώντας με ένα προϋπολογισμό ένα έτος, να δει κατά πόσο επαρκεί το προσωπικό της και αν όχι, αν διαπιστώσει πως δεν επαρκεί, μπορεί να υποβάλει συμπληρωματικό προπολογισμό και μπορεί και κατά τη διάρκεια του έτους ε, προπολογισμού, του οικονομικού έτους, να υπάρξει μία τροποποίηση του ήδη εγκεκριμένου προπολογισμού. Αυτά σε ό,τι αφορά τι υπηρεσίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα νέα ε, ποσά του προπολογισμού. Προφανώς και ακούγεται πολύ ωραίο το να προσπαθήσει κανείς να δημιουργήσει νέα σημεία στον προπολογισμό, νέα κονδύλια και να λέει πως υπάρχει πολιτική βούληση για αυτό το σημείο. Πολύ καλά λοιπόν καταγράφει κανείς έτσι την πολιτική του βούληση, αλλά αυτό δεν μας βοηθάει γιατί προϋπολογισμός και γραμμές προϋπολογισμού μπορούν να προκύψουν μόνο με βάση συγκεκριμένη νομική βάση και η Επιτροπή η οποία καλείται να εκτελέσει αυτό το προϋπολογισμό χρειάζεται συγκεκριμένη νομική βάση ε, επί τη βάση της οποίας θα ε, γίνει η εν λόγω δαπάνη. Πέρυσι οι συνάδελφοί μου δεν ήθελαν να με ακούσουν. Είχαμε για παράδειγμα μια γραμμή του προπολογισμού για το κλίμα. Γιατί δεν με ακούνε οι συνάδελφοι. Και αυτά τα 20 εκατομμύρια ευρώ τα οποία έχουν μπει σε αυτή τη γραμμή του προπολογισμού δεν είναι δυνατόν να δαπανηθούν. Δεν μπορεί να τα δαπανήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσπαθεί να δει πώ μπορεί να μεταθέσει αυτά τα κονδύλια σε άλλε γραμμέ του προπολογισμού και να μπορέσει να τα δαπανήσει. Άρα λοιπόν ε, αυτό είναι ανόητο που κάνουμε. Ουσιαστικά βάζουμε κάπου ε, κονδύλια και τελικά δεν μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε επειδή δεν υπάρχει νομική βάση για την ε, αξιοποίησή τους. Α μην δημιουργούμε έτσι απλά γραμμέ του προπολογισμού. Α είμαστε πιο προσεκτικοί, α εξετάσουμε τι ε, συγκεκριμένε γραμμέ που υπάρχουν και α πούμε εδώ θέλουμε να δώσουμε περισσότερη έμφαση. Εκεί θέλουμε να δαπανίσουμε περισσότερα κονδύλια. Όλα τα άλλα όχι. Τρίτο σημείο. Πιλωτικά προγράμματα. Οι συνάδελφοι Ε, ήταν ε, ε, πέτυχαν, δεν θα το έλεγα πέτυχαν, εν πάση περιπτώσει ήταν πολύ εφευρετικοί σε ό,τι αφορά τα πιλωτικά προγράμματα. Πολλές από τις προτάσεις για τα πιλωτικά προγράμματα τελικά αποσύρθηκαν, αλλά όχι όλες. Υπήρξαν δηλαδή κάποιες που παρέμειναν. Να σας υπενθυμίσω πως τα πολιτικά προγράμματα και οι, τα προπαρασκευαστικά έργα καταρχήν θα πρέπει να πληρούν ένα κριτήριο, να έχουν ευρωπαϊκή υπεραξία επιπρόσθετη δηλαδή χρησιμότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι καινοτόμα, πραγματικά ρηξικέλευτα. Δεν μπορεί να ε, υπάρξει, υπάρχει ήδη κάποια άλλη νομοθεσία ή κάποιο άλλο πρόγραμμα το οποίο καλύπτει ε, τα εν λόγω ε, ζητήματα. Μπορεί να πρόκειται για μια καλή, μια σωστή πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου, αλλά δεν αποτελεί σε αυτή την περίπτωση πιλωτικό πρόγραμμα. Άρα και γι' αυτό θα πρέπει να πω δυστυχώ στον κύριο Ζέμπερ πω τα δύο προτινόμενα από την τρίτη πλευρά πιλωτικά προγράμματα δεν αποτελούν πιλωτικά προγράμματα. Δεν είναι καινοτόμα. Το ίδιο ισχύει και για τον συνάδελφο που κάθεται δίπλα μου τον κύριο Άντερ. Δηλαδή να έχουμε ένα συγκεκριμένο πιλωτικό πρόγραμμα περιφερειακό, αλλά ήδη έχουμε, ε, ακόμα και με 11 κράτη-μέλη τα οποία συμμετέχουν σε αντίστοιχο πιλωτικό πρόγραμμα. Και θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να, να προτείνουμε κάτι αντίστοιχο για διεύρυνση ενδεχομένω του προγράμματο, αλλά δεν μπορούμε να προτείνουμε ε, ε, άλλο τέτοιο εναλλακτικό πρόγραμμα. Και για, ε, στο Chris θα ήθελα να πω ότι με αυτή την καλή ιδέα ε, το, την ε, καλλιέργεια, δηλαδή τις καλλιέργειες με, χαμηλή, με χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα έχει καθυστερήσει κατά περίπου 9 μήνες. Δηλαδή ήδη υπάρχει μια μελέτη που έχει εκμονηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, τα αποτελέσματα θα τα λάβουμε εμείς αρχές του ερχόμενου έτους. Άρα και εδώ λοιπόν μας έχει προλάβει ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιλωτικό πρόγραμμα δεν μπορεί εδώ να γίνεται λόγος ότι πράγματι αποτελεί αυτή η πρόταση. Ε, του κυρίου Τόμας ε, Ούλμα, ε, η πρόταση για το πρόγραμμα δηλαδή για την υπατήτητα Β, ναι, εκεί πραγματικά έχουμε να κάνουμε πιλωτικό, δηλαδή καινοτόμο πρόγραμμα και μπορούμε να το εγκρίνουμε. Αυτά από την πλευρά μου. Ευχαριστώ, ε, Κιούτα ήταν πολύ χρήσιμο το ότι μας εξήγησε σε μία ακόμα φορά το πώς έχουν τα πράγματα σε σχέση με τις υπηρεσίες και με τις γραμμές του προπολογισμού. τώρα θα ήθελα να ζητήσω την κατανόησή σας γιατί έχουμε δύο προέδρους του Συμβουλίου σε 10 λεπτά που θα είναι εδώ μαζί μα ε, και τώρα έχουμε τόσο λίγο χρόνο για να εγκρίνουμε τον προπολογισμό. Πάντα συμβαίνει αυτό, δηλαδή ω ε, νέο κοινοβούλιο να μην έχουμε εκ των προτέρων χρόνο στη διάθεσή μα για να συζητήσουμε μετά τον προπολογισμό. Δυστυχώ έτσι έχουν τα πράγματα, οπότε θα ήθελα να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία και ε, ζητώ την κατανόηση των συναδέλφων οι οποίοι θα ήθελαν να πούν κάτι, αλλά βέβαια ο καθένα έτσι αλλιώ μπορεί να αποφασίσει όπω αυτό θεωρεί. Ε, περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία στη πρώτη τροπολογία 5911, η ψήφη υπέρ. Ηλεκτρονικά, λέει ο πρώτος, όχι. Ε, ψήφι κατά, αποχές, κρίνεται. 5905, η Γιούτα Χάουγκ, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, εκρίνεται. 5910, Γιούτα Χάουγκ, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 59-21, Chris Davis, ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές. Θα πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψήφι υπέρ. Ζητώ συγγνώμη, λέει η Γιώτα Χάουγκ. Εδώ δεν έχουμε καθόλου να κάνουμε με το πιλωτικό πρόγραμμα του Κριστέβης. Ε, οι τροπολογίε 59-21 και 59-13 είναι ουσιαστικά ταυτόσιμε. Πρόκειται δηλαδή για μια αλλαγή σε ό,τι αφορά την γραμμή του προπολογισμού 07-03-07. Είναι ταυτόσιμε. Καλώ. Ε, ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. ...35 ψήφοι υπέρ, 0 κατά, μία αποχή, άρα εγκρίνεται. Κρίς, θέλεις το λόγο. Ναι. Έχουν, τουλάχιστον δύο συνάδελφοί μου εδώ έχουν τρεις τέσσερις, τέσσερις συνάδελφοι των οποίων τα μηχανήματα δεν λειτουργούν, έτσι. Άρα χαιρόμαστε με αυτό το αποτέλεσμα, γιατί σίγουρα δεν θα είχε αλλάξει το τελικό αποτέλεσμα, αλλά εν πάση περιπτώσει να δούμε πώς ε, μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τα μηχανήματα ψηφοφορίας. Μετά ε, πρέπει να ψηφίσουμε και επί της 5906. Γιούτα Χάουκ. Ψήφι υπέρ της τροπολογίας 5906. Ψήφι κατά. Αποχές εγκρίνεται. τέσσερα Μας Ε, το λόγο. Ναι, είχα προτείνει αρχικά στον ΠΑΣ να μεταφερθούν τα όσα πρότεινε, αλλά αφού ε, το συζητήσαμε, ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε πως μπορεί να το εφαρμόσει και μέσα στο ε, Life Sin, Life Plus. Γιατί συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το πρόγραμμα, οπότε μπορούμε να ψηφίσουμε ε, επ' τη τροπολογία τροπολογίας ε, του Μπα, ω έχει χωρίς δηλαδή προφορική τροποποίηση της από τη ΧΑΟΚ ψηφι Ψήφι υπέρ λοιπόν. Ψήφι κατά. Αποχές εγκρίνεται. 59-14 Γιάννο Άντερ. Ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές εγκρίνεται. 59-18, Ρίχαρτ Ζίμπερ. Ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 59-19, Ρίχαρτ Ζέμπερ. Ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές. Μπορούσε να είναι το 50-50 τι θα κάνουμε τώρα με τα μηχανήματα που δεν λειτουργούν. Α δοκιμάσουμε ξανά για τι ηλεκτρονική οδού και μετά όσοι, όσον τα μηχανήματα δεν λειτουργούν θα πρέπει να του τους προσμετρήσουμε ανάταση χειρός. Ψηφίζουμε επί τη 59-19, τη ψηφοφορία λοιπόν. «43 ψήφισαν, 20 υπέρ, 22 κατά, μία εποχή. Θα πρέπει να μετρήσουμε. Ζητώ συγγνώμη. Πρέπει να μετρήσουμε γιατί υπάρχουν πολλά μηχανήματα που δεν λειτουργούν. Ζητώ από τη γραμματεία να καταμετρήσει λοιπόν τις ψήφους. 59-19 ψήφοι υπέρ της 59-19 του Ρίχαρτ Σέμπερ.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 26 υπέρ 32 κατά ζητώ συγγνώμη Ρίχαρτ απορρίφθηκε 59-20 Chris Davis ψήφι υπέρ ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται 59-26 Utah Hawk ψήφι υπέρ ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται 59-15 Έχουμε δύο ταυτόσημες, 59-15 και 59-16. Ψήφι υπέρ. Α, όχι, έχουμε ξεχωριστή ψηφοφορία, split vote. Για το πρώτο τμήμα λοιπόν ψηφίζουμε. ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5908 Γιούτα Hawks ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5909 Γιούτα Hawks ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5924 Τόμας Ούλμαρ ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. εποχές θα πρέπει να μετρήσουμε Ψήφι υπέρ λοιπόν ξανά. Για την 59-24 του Τόμας Ούλμερ. Ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. 30 υπέρ προς 20 κατά, άρα εγκρίνεται. 5907 Γιούτα Χάουκ. Ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές εγκρίνεται. 59-12. Γιούτα Χάουκ. Ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5925 Τόμας Ούλμερ, ψήφι υπέρ, ψήφι κατά, αποχές εγκρίνεται και 5903 Μπας Άικουτ Γιούντις Αργεντίνη, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ολοκληρώσαμε με αυτή την ψηφοφορία. Σε ευχαριστούμε Κιούτα Χάουγκ για τη δουλειά σου εδώ και σας ευχαριστώ όλους για την κατανόησή σας για αυτήν την κάπως εξαιρετική διαδικασία που ακολουθήσαμε.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 So, liebe Αγαπητοί κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, ε, περνάμε στο επόμενο σημείο τη ημερή σα διάταξη. Ε, καλωσορίζω λοιπόν θερμά. Σα παρακαλώ λίγο την προσοχή σα. Ξέρω πω έχετε πολλά να συζητήσετε, αλλά συγκεντρωθείτε λίγο. Ντάγμαρ, θέλουμε να συνεχίσουμε. Σα παρακαλώ. Hello. Okay. Now we can start. Yeah. Uh... Ωραία. Μπορούμε λοιπόν να αρχίσουμε. Καλωσορίζουμε λοιπόν ε, θερμά εδώ τη Σουδική Προεδρία, εκπροσώπους εδώ, δύο εκπροσώπους μαζί, δύο σε έναν εκπροσώπους και χθε είχαμε εκπροσώπους από τη Σουδική Προεδρία. Σήμερα έχουμε λοιπόν μαζί μας τον κύριο Γκέραν Χέγκλουντ, Σουδηδό Υπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας και την κυρία Μαρία Λάρσον, στον Υπουργό Τρίτη Ηλικίας και Δημόσιας Υγεία. Α χειροκροτήσουμε λοιπόν εδώ τους δύο υπουργού που βρίσκονται σήμερα εδώ μαζί μας στην Επιτροπή μας. Γνωρίζουμε πως ε, η Σουηδική Προεδρία είναι πολύ φιλόδοξη, πολύ καλά προετοιμασμένη. Ήδη λάβαμε κάποια γεύση από το έργο σας ε, μέσα σε αυτή τη βδομάδα, από τις παρουσιάσεις σας ε, και αναμένουμε τώρα με μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια να ακούσουμε τα όσα έχει να μας πείτε εσείς ως προς τα όσα θέλετε να κάνετε στα δικά σας, στους δικούς σας ε, τομείς. Οπότε χωρίς να χάνουμε περαιτέρω χρόνο να δώσω το λόγο στον κύριο Γκέραν Χέγγλουμ. Παρακαλώ. Χίλια ευχαριστώ Πρόεδρε για τα θερμά σας λόγια. Μας καλωσορίσατε και οι σχέσεις που οικοδομούμε σήμερα θα διαδραματίσουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ούτως ώστε να προάγουμε διάφορα σημαντικά ζητήματα μέσα από την συνεργασία μας. Με τιμά ιδιαίτερα που έχω την ευκαιρία σήμερα να παρευρεθώ συνεδρία της Επιτροπή Περιβάλλοντος για να συζητήσουμε μαζί τα ζητήματα της υγείας και πώς θα εξελιχθούν υπό Σουηδική ε, Προεδρίας. Θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ τυχερός ε, που μπορώ να ασχολούμαι με θέματα υγείας γιατί η υγεία έχει ζωτική σημασία στην καθημερινή ζωή όλων των ανθρώπων. Ε, και το ίδιο ισχύει και για τους συγγενείς και για τους συμπολίτε μας. Την ε, περασμένη άνοιξη, πριν από τις εκλογές του Κοινοβουλίου, το Ευρωβαρόμετρο έδειξε ότι τα θέματα τα, των, της προστασίας των καταναλωτών και της προστασίας ε, της υγείας έχουν την μεγαλύτερη σημασία, το μεγαλύτερο ειδικό βάρος. Το ίδιο και η απασχόληση. Είναι κοινή μας ευθύνη λοιπόν να ασχοληθούμε με όλα αυτά τα σημαντικά για τους συμπολίτες μας ε, ζητήματα και συνιστά αυτό μεγάλη πρόκληση για τα επόμενα πέντε χρόνια. Ε, ο στόχος μας είναι οι πολίτες ε, να μπορούν να έχουν την βέλτιστη δυνατή υγειονομική περίθαλψη όταν ε, την χρειάζονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μας προσφέρει μια καλύτερη υγεία. Βέβαια είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι μεγάλο μέρος της ευθύνης ανήκει στα κράτη-μέλη για τα θέματα υγείας. Υπάρχουν περιορισμοί ως προς τις πρωτοβουλίες που μπορούν να ληφθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλα αυτά, παρά την εθνική ευθύνη, παρά τις προκλήσεις, οι οποίες καλούνται να τα τα κράτη-μέλη, θεωρούν ότι μπορούμε να μάθουμε πολλά ο ένας από τον άλλον μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον τομέα της υγείας και για τους συμπολίτε μας υπάρχει μια σαφής προστιθέμενη αξία που θα προκύψει από την, συνεργασία, την διακρατική συνεργασία Σήμερα θα συζητήσουμε διάφορα ζητήματα ε, και για όλα αυτά ε, η ικανότητα του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου να συνεργαστούν και να συμφωνήσουν θα είναι η προϋπόθεση για να ληφθούν οι αποφάσεις που θα αποσκοπούν στο να αναβαθμιστεί η κατάσταση για τους ασθενείς στην Ευρώπη. Μιλάμε, Φερρυπίνη, για την οδηγία για τα δικαιώματα των ασθενών, για αποζημίωση όταν λαμβάνουν περίθαλψη σε κάποια άλλη χώρα και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουν ναι, οι επικοδομητικές συζητήσεις για αυτό το θέμα το φθινόπερο και θέλω πραγματικά να τονίσω πόσο σημαντικό είναι για μας ε, να τονίσω τη βούλησή μας ε, να έχουμε μια αγαστή συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Είναι, συμφέρον, είναι προς το δικό μας το συμφέρον, προς το δικό σας συμφέρον και κυρίως και πάνω απ' όλα προς το συμφέρον των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταφέρουμε να συνεργαστούμε με επικοδομητικό τρόπο να επιφέρουμε τι απαιτούμενε κατά τη γνώμη μα βελτιώσει στον τομέα τη υγεία. Θα ήθελα τώρα, εν συντομία, να σα παρουσιάσω τα θέματα που επέλεξε η Σουηδική Προεδρία να ε, ιεραρχίζει ως προτεραιότητες κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου. Στον τομέα, εγώ είμαι αρμόδιος για τα θέματα υγείας και υγειονομικής περίθαλψης και η συνάδελφός μου, η Μαρία Λάρσον, ασχολείται με τα θέματα δημόσιας υγείας. Γι' αυτό θα ακούσετε δύο παρουσιάσεις. Το φθινόπωρο θα είναι εντατικότατε οι εργασίε μα. Έχουμε πάρα πολλά ζητήματα στην ημερήσια διάταξη και δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Αυτό σημαίνει μια μεγάλη πρόκληση για την Σουηδική Προεδρία. Παρόλα αυτά θα σπεύσουμε βραδέως. Ε, θα είμαστε προσεκτικοί γιατί υπάρχουν πολλές καλές δυνάμεις εισαγωγικά που μπορούν να συνεργαστούν και ξέρουμε ότι μόνοι μας δεν πρόκειται να τα καταφέρουμε. Οπωσδήποτε πρέπει να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη, με το Κοινοβούλιο και φυσικά και με την Επιτροπή, ούτω ώστε να ευοδοθούν οι προσπάθειές μας. Ε, θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο να ε, εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να ευχαριστήσω και τους Γάλλους και Τσέχους συναδέλφους μου για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε στο παρελθόν. Η δουλειά που έκαναν τον περασμένο χρόνο, κυρίως ως προς την οδηγία για τα δικαιώματα των ασθενών και το θέμα της ε, αντοχής στα αντιβιωτικά, η εργασία τους λοιπόν συνέβαλε με καταλητικό τρόπο και μας έδωσε την ε, ευκαιρία ε, να μπορούμε να ελπίζουμε κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου να καταλήξουμε σε μια πολιτική συμφωνία. Και ακόμη και η επερχόμενη Προεδρία, η Ισπανική, ε, θα συνεργαστεί μαζί μας για να υπάρχει και η απαιτούμενη συνέχεια στις εργασίες του Συμβουλίου. Η Προεδρία μας άρχισε, όπως γνωρίζετε, το, την 1η Ιουλίου με ιδιαίτερη δυναμικότητα, αν θέλετε, γιατί ήδη στο Gen Shopping στις 6 και 7 Ιουλίου οργανώσαμε ένα άτυπο Συμβούλιο Υπουργών. Εκεί συζητήσαμε την οδηγία για, τις, για τα δικαιώματα των ασθενών, ε, ρίχνοντας βάρος όλος ιδιαίτερος στις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκεί ε, συζητήθηκαν οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου που υπευλήθησαν στην πρώτη ανάγνωση, ούτω ώστε όλα τα κράτη-μέλη να ενημερωθούν για τη θέση του Κοινοβουλίου και συζητήσαμε για το ποιε θα μπορούσαν να είναι μελλοντικέ μας κινήσει. Και οι υπουργοί υπέδειξαν ποια είναι τα σημαντικά ζητήματα για κάθε μία χώρα για τις μελλοντικέ συζητήσεις. Ε, και στο αυτό το άτυπο συμβούλιο συζητήσαμε το θέμα της αντίστασης ε, στο αντιβιωτικά του αλκοόλ και των αλκοολούχων ποτών και της νέας γρήπη. Ε, το πρώτο βασικό συμβούλιο θα γίνει το Δεκέμβριο στις Βρυξέλλες, παρότι θα έχουμε για το θέμα της γρήπης ένα έκτακτο συμβούλιο στις 12 Οκτωβρίου και θα συνεχίσουμε να διοργανώνουμε διάφορες διασκέψεις εμπειρογνωμόνων για, για μια σειρά ζητημάτων και σε ορισμένες από αυτές τις διασκέψεις θα καλέσουμε και υπουργού και βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλουμε πραγματικά να είναι ενεργός η εμπλοκή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην όλη διαδικασία, ούτω ώστε να μπορέσετε ήδη σε αρχικό στάδιο να επηρεάσετε τη διαδικασία ε, διαμόρφωσης της νομοθεσίας και τη της μελλοντικής κοινή πολιτικής στον τομέα αυτό. Θα ήθελα τώρα να εξετάσω διεξοδικότερα κάποια ζητήματα που θα μας απασχολήσουν. Πρώτον, οδηγία για το δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης σε άλλη χώρα για τους ασθενείς. Ε, σας είπα ήδη κάποια πράγματα. Ξέρετε ότι από πολιτική σκοπιά είναι δύσκολο το θέμα. Υπάρχουν, υπάρχει μεγάλη διάσταση απόψεων ανάμεσα στα κράτη-μέλη και ε, το Κοινοβούλιο έχει εκφράσει σαφώς επιθυμίες του σε αυτό το τομέα τομέα. όπω σα είπα, η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια οδηγία για τα δικαιώματα των ασθενών για περίθαλψη σε άλλη χώρα συζητήθηκε ήδη υπό Γαλλική και Τσεχικής Προεδρίας. Η οδηγία έχει ως στόχο αρχικά να διευκρινίσει την ομολογία του 10 στον τομέα αυτό και οι συζητήσει στο Συμβούλιο εστιάζουν ως επιτοπλίστων στο να βρεθεί μια ισορροπία ε, ανάμεσα στα δικαιώματα των ασθενών αφενός για διασυνοριακή περίθαλψη και ε, την ευθύνη των κρατών μελών αφετέρου για να οργανώσουν την, ε, τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και, κοινωνικής, και υγειονομικής περίθαλψης. Συγγνώμη και φυσικά έχουμε λάβει υπόψη τη γνωμοδότηση για αυτό το θέμα του Κοινοβουλίου. Έχουμε ως στόχο να καταλήξουμε σε πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο το φθινόπερο, αλλά αυτό βέβαια είναι συνάρτηση της Βούλης των κρατών μελών να συνεχίσουν τις επικοδομητικές συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις για να καταλήξουμε σε συμβαστική λύση, παρότι έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα και έχει σημειωθεί πρόοδο, εκκρεμούν διάφορα ζητήματα. Παραδείγματο χάρη, το πεδίο εφαρμογή αυτή τη οδηγία, κυρίω ω προ ε, του ιδιωτικού φορεί υγειονομική περίθαλψη, ε, που δεν ε, καλύπτονται από το σύστημα κοινωνική ασφάλιση στη χώρα υποδοχή και μηχανισμοί για συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη ω προ το κεφάλαιο 4 τη οδηγία για τα θέματα κοινωνική πρόνοια και κοινωνική ασφάλιση. Επίση, πρέπει να διασφαλίσουμε ένα εύλογο επίπεδο ασφάλεια και ποιότητα για τη διασυνοριακή περίθαλψη. μεγάλε οι προκλήσει. Ελπίζω να έχει οριμάσει ο καιρό τόσο ώστε να καταλήξουμε το φθινόπωρο σε πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο και ε, υπολογίζουμε στην ε, πλήρη υποστήριξη και του Κοινοβουλίου και τη Επιτροπή και του Συμβουλίου για να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Είναι μεγάλη φιλοδοξία μας ε, και μια κοινή θέση θα αποτελέσει μια καλή βάση για μια επικοδομητική δεύτερη ανάγνωση. Α περάσουμε στο πακέτο των φαρμάκων ένα άλλο ευρύτατο θέμα που ε, σκοπεύουν να εξετάσουμε είναι οι νομικές πράξεις για το πακέτο των φαρμάκων ναι, που αποτελείται από τρία τμήματα. Ε, ενημέρωση του κοινού, ε, παραποιημένα ή ψευδεπίγραφα φάρμακα και τέλος φαρμακοεπαγρύπνηση. Θα ήθελα να αρχίσω με το πλέον ευαίσθητο κομμάτι του πακέτου, δηλαδή με τις πληροφορίες για τα φάρμακα προς το κοινό. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας έκδηλα προέκυψε ότι πολλά κράτη-μέλη θέλουν να αποδώσουν ύψιστη προτεραιότητα στα άλλα δύο τμήματα του πακέτου, δηλαδή τα παραποιημένα φάρμακα και την φαρμακοεπαγρύπνηση. Αυτό είναι μια προσέγγιση που και εμείς συμμεριζόμαστε από πλευράς μας, ε, διότι Προ το παρόν δεν πρόκειται να συνεχίσουμε τι διαπραγματεύσει στο Συμβούλιο. Προέβαλε ενστάσει στο Συμβούλιο για την δυσδιάκριτη συνοριακή γραμμή ανάμεσα στι διαφημίσει και τι πληροφορίε για τα φάρμακα, το ρόλο τη φαρμακοβιομηχανία και εξάλλου πολλά κράτη-μέλη έχουν και ενστάσει συνταγματικού χαρακτήρα που σίγουρα δύσκολα θα υπερπηδηθούν. Τώρα το φθινόπωρο αποφάσισε το Συμβούλιο να αφιερώσει το χρόνο του στα άλλα δύο κομμάτια του πακέτου των φαρμάκων. Παραδείγμα, για το, τα παραποιημένα φάρμακα ε, τον περασμένο χρόνο ε, παρατηρήθηκε ότι πέρασαν ε, μεγάλα, πάρα πολλά παραποιημένα φάρμακα μέσα στην νόμιμη αλυσίδα διανομής και θέλουμε αυτό να το παρεμποδίσουμε μέσα από αυτή την πρόταση. Επίσης, για την φαρμακοεπαγρύπνηση θα θέλαμε να γίνει πιο αποτελεσματική η προστασία και να καταστεί σαφές ποιος θα έχει την ευθύνη για την υποβολή εκθέσεων για τις παρενέργειες των φαρμάκων στην Ευρώπη. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προχωρήσει η διαδικασία και ελπίζουμε με το που θα αρχίσουν εργασίες στο Κοινοβούλιο ουσιαστικά να εντατικοποιηθεί η συνεργασία ανάμεσά μας. Ε, θέλουμε να συνεργαστούμε με τους νέους εισηγητές για αυτά τα θέματα ε, μόλις διοριστούν για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία το ταχύτερο δυνατόν. Το επόμενο θέμα που θέλω να σχολιάσω είναι η αντοχή στα αντιβιωτικά και το... η ηλεκτρονική υγεία. Ε, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας έχω αναλάβει πρωτοβουλία για συμπεράσματα συμβουλίου για δύο σημαντικούς τομείς. Ε, αντοχή στα αντιβιωτικά και η ηλεκτρονική αγία. Αυτή η αντοχή στα αντιβιωτικά είναι μια πολύ σοβαρή απειλή για το μέλλον και πρέπει οπωσδήποτε να ασχοληθούμε με την υγιεινή στους χώρους παροχής περίθαλψης ε, και με την μείωση της εθνικής συνταγογράφησης. Υπάρχει όμως και ένας τομέας ε, που συχνά παραλείπουμε στις συζητήσεις μας, συγκεκριμένα έρευνα και ανάπτυξη νέων αντιβιωτικών. Σήμερα δεν υπάρχουν επαρκή κίνητρα για να γίνει η έρευνα για νέα φάρμακα νέα φάρμακα που χρειαζόμαστε και ως εκ τούτου προέκυψε ένα χάσμα ανάμεσα στην ανάγκη για τα νέα αντιβιωτικά και τις τωρινές εξελίξεις ε, αυτών των, ε, την τωρινή ανάπτυξη αυτών των φαρμάκων. Χρειαζόμαστε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή θεσμοί και η φαρμακοβιομηχανία για να βρούμε νέες λύσεις. Χρειαζόμαστε μια νέα γενιά αντιβιωτικών ε, για να καλύψουν το κενό και τις ατέλειες των αντιβιωτικών που ε, ήδη υπάρχουν και φυσικά η διεθνής διάσταση έχει ιδιαίτερη σημασία. Γίνει δηλαδή μια διεθνής προσπάθεια. Τώρα, για την ηλεκτρονική υγεία θέλουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να τονίσουμε τη σημασία της ηλεκτρονικής υγείας ε, στην ε, πολιτική ημερήσια διάταξη. Δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα νέα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας από την πληροφορική, ούτως ώστε η υγειονομική περιθέλψη και η κοινωνική πρόνοια να, είναι, ε, ε, να γίνονται με ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο τρόπο. Και έχουν γίνει υπολογισμοί που δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλο δυναμικό ανάπτυξη αν χρησιμοποιήσουμε τα νέα εργαλεία. Δηλαδή θα υπάρχει καλύτερη σχέση κόστους-οφέλους για τους πολίτες και θα είναι καλύτερη η περίθαλψη ε, για όλους όσους την χρειάζονται. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ε, στα πλαίσια μιας ε, ενδεχόμενης συμφωνίας σε αυτό το τομέα. Τέλος, ας αναφερθώ παρόδο στη δωρεά οργάνων και στις μεταμοσχεύσεις. Θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις υπό την Προεδρία μας με τα κράτη-μέλη αλλά δεν πρόκειται να έχουμε αρκετό χρόνο ώστε να καταλήξουμε σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Θα το αφήσουμε για την Ισπανική Προεδρία. Ιδού, αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα και πάλι πριν κλείσω να τονίσω πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μια στενότατη συνεργασία για να επιτύχουμε όλους αυτούς τους κοινού μας στόχους και θα δώσω το λόγο στην Υπουργό Μαρία Λάρσον και ελπίζω ότι μετά θα γίνει μια ε, επικοδομητική συζήτηση και το φθινόπωρο θα έχουμε όλοι μια αγαστή συνεργασία όπως σας έλεγα. Πρόεδρε, Αξιότιμοι βουλευτές, θα ήθελα να συμφωνήσω με τα τελευταία λόγια του Γέραν Χέγκλουντ. Ε, δηλαδή, χαίρομαι πάρα πολύ που έχω την ευκαιρία να σας συναντήσω σήμερα και εύχομαι ε, να αποτελέσει η σημερινή μας συνάντηση τη βάση μιας πολύ καλής συνεργασίας το φινόπορο. Θα ήθελα να συγχαρώ τους νεοεκλεχθείς ε, που αρχή, κυρίως αυτούς που έχουν την πρώτη τους ε, θητεία και να τους ευχηθώ καλή επιτυχία λοιπόν για τις εργασίες εργασίες τους. Εγώ ασχολούμαι με θέματα δημόσιας υγείας και μπορούμε να πούμε ότι χρειάζονται συντονισμένες παρεμβάσεις και μια συνεργασία για τα θέματα δημόσιας υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η ανάγκη είναι όλο ένα και πιο επίκαιρη. Πολλά, πολλές από τις προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι κοινέ στην Ευρώπη παρατηρούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη και άρα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε από κοινού. Για, επίσης, σε καμία χώρα δεν πρόκειται να γλιτώσει από τις επιπτώσεις ε, της νέας γρήπης HNN1. Ε, και βλέπουμε πόσο μεγάλη σημασία έχουν υπάρχουν οι πανδημίες ε, και πόσο σημαντικό είναι να είμαστε καλά προετοιμασμένοι σε εθνικό επίπεδο, σε κοινοτικό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα ήθελα αρχικά να σας μιλήσω για τις παρεμβάσεις μας στον τομέα της καταπολέμησης αυτής της πανδημίας και μετά θα αναφερθώ σε κάποια άλλα ζητήματα δημόσιας υγείας που θα αναδείξουμε σε προτεραιότητες κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Τα κράτη-μέλη ε, επί σειρά ετών ε, προετοιμάζονταν για την πανδημία γρήπη το 2005 συγκροτήθηκε το ECDC που είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Προστασία κατά των μεταδοτικών ασθενειών στην ε, Στοκχόλμη έχει την έδρα του και αυτή η αρχή έχει επικουρήσει τα κράτη-μέλη ε, με πάρα πολύ αξιόλογες γνώσεις και καλή επιστημονική βάση για να αντιμετωπιστεί το θέμα της γρήπης. Ε, και σας, γι' αυτό σας είπα, χάρη αυτό, και σε αυτό το κέντρο είμαστε καλά προετοιμασμένοι σήμερα σήμερα. Το 2007 αποφάσισε το ECDC ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση ετοιμότητας ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ότι έπρεπε να αναπτυχθούν περαιτέρω κάποια, ε, κάποια μέτρα. Ε, έκτοτε όντως αναλύθηκαν και άλλα μέτρα και εδώ και χρόνια συζητούμε αυτό το θέμα αφιέρωσαν, ε, αφιερώθηκαν πάρα πολλά ε, ε, υπουργικά συμβούλια σε αυτό το θέμα για να δούμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να αντιμετωπίσουμε τις επιβλαβείς συνέπειες μιας ενδεχόμενης κρίσης. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ένας ακρογωνίος λίθος της διεθνούς συνεργασίας είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αλλά και οι παρεμβάσεις που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνονται και υπό την αιγίδα του ΠΟΕ αλλά και ε, σύμφωνα με τις ε, διατάξεις του ΠΟΕ θεωρώ ότι μπορούμε να βελτιώσουμε το συντονισμό σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και να προετοιμαστούμε. Παρότι υπάρχει καλό επίπεδο ετοιμότητα, αλλά πάντοτε μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Οι εργασίε άρχισαν υπό Τσεχική Προεδρία. Ε, συγκάλεσε η τσεχική προεδρία 30 Απριλίου ένα έκτακτο υπουργικό συμβούλιο και σίγουρα θα συνεχίσουμε αυτέ τι εργασίε. Στο άτυπο υπουργικό συμβούλιο στο Γιάνν Σέπινγκ που έγινε στι αρχέ του Ιουλίου συζητήθηκε η γρήπη και πολλοί εξέφρασαν την υποστήριξή τους ε, για την ενδεχόμενη υιοθέτηση συμπερασμάτων από το Συμβούλιο το φθινόπωρο που για ε, θέματα με στρατηγική σημασία για τη μελλοντική μας συνεργασία. Και ε, ένα έκτακτο Συμβούλιο θα συγκαλέσουμε στις 12 Οκτωβρίου για να συζητήσουμε το θέμα της, γρήπ, της γρήπης συγγνώμη, και να ευελπιστούμε ότι εκεί θα υιοθετηθούν και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Στα πλαίσια των συνθέσεων του Συμβουλίου, εμείς επανεργοποιήσαμε το, την ομάδα των φίλων της Προεδρίας για τα θέματα της γρήπης, για να αντιμετωπίσουμε την κρίση και να δούμε ε, ποια ποιες είναι οι πολυτομιακές ε, διαστάσεις αυτής της πανδημίας. Ε, κάποια ζητήματα που θα εξετάσουμε το φθινόπωρο είναι μεταξύ άλλων πρόσβαση στα εμβόλια, δυνατότητα κοινή διαχείρισης των εμβολίων για τα κράτη-μέλη που σήμερα ε, δεν έχουν συμβάσεις ε, με την φαρμακοβιομηχανία για την παράδοση εμβολίων. Ε, παγκόσμια αλληλεγγύη, κάποια κοινή επικοινωνιακή πολιτική και πολυτομιακά ζητήματα τα οποία πρέπει να επεξεργαστούμε περαιτέρω αλλά από σκοπιάς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το παρόν εργάζεται εντατικά για αυτό το θέμα της γρήπης ε, και η πρόθεσή τους είναι να εκδώσουν ανακοίνωση ε, στα μέσα Σεπτεμβρίου για αυτό το θέμα. Θα θεωρούμε ότι αυτό θα αποτελέσει πάρα πολύ σημαντικό βήμα για τις εργασίες ε, της ομάδας των φίλων της Προεδρίας στο Συμβούλιο και για το Υπουργικό Συμβούλιο που θα λάβει η χώρα στις 12 Οκτωβρίου. Ε, κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστεί να επανέλθουμε σε διάφορα βήματα σε αυτό το θέμα κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου και ελπίζω να δείξετε κι εσείς ε, αντίστοιχη προσήλωση και δέσμευση για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Τον Ιούλιο επίσης εκδόθηκε σύσταση σε σχέση με τον εμβολιασμό της ετήσιας γρήπης αυτής που μας ε, πλήττει κάθε χρόνο δηλαδή. Προβλέπονται εθνικά σχέδια δράσης για να εκπληρωθεί ο στόχος σε συγκεκριμένα ο εμβολιασμό του 75% των ατόμων που υπερβαίνουν τα 65 χρόνια. Η Σουηδική Προεδρία θα αρχίσει τις διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο για αυτή την σύσταση περί εμβολιασμού. Θα ήθελα τώρα να περάσω σε κάποια άλλα επίκαιρα ζητήματα. Πρώτον, αλκοόλ θα γνωρίζετε κατά πάσα πιθανότητα ότι στην πρώτη μας Προεδρία το 2001 οργανώσαμε μια ενισχυμένη συνεργασία ανάμεσα ε, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μειώσουμε τις επιβλαβείς επιπτώσεις ε, του αλκοόλ. Ε, υιοθετήθηκε κοινή στρατηγική στον τομέα αυτό και θέλουμε να δώσουμε μια συνέχεια σε αυτή την πολύ σημαντική εργασία που έγινε το 2001. Το φθινόπωρο Έχουμε ήδη προβλέψει σε στενή συνεργασία με τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΣΑΝΚΟ και μια παγκόσμια διάσκεψη εμπειρογνωμόνων και μια ευρωπαϊκή διάσκεψη εμπειρογνωμόνων και ελπίζουμε να εγκριθούν συμπεράσματα από το Συμβούλιο για το αλκοόλ και τις επιπτώσεις στην υγεία το Δεκέμβριο. Αναμένουμε τα συμπεράσματα να εστιαστούν στους νέους και το αλκοόλ, ε, στην θέση σε εμπορία και στις ε, γενικότερες βλαβερές συνέπειες του αλκοόλ. Ε, στην παγκόσμια διάσκεψη εμπειρογνωμόνων ε, θα δώσουμε το βάρος στη σχέση ανάμεσα στο αλκοόλ, τη φτώχεια και την ε, διάδοση των μεταδοτικών ασθενειών σε χώρες χαμηλού και μέσου εισοδήματος. Αυτό θα το διοργανώσουμε σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Επίσης, να αναφερθώ και σε μια διάσκεψη που ε, θα γίνει εδώ στο Κοινοβούλιο την άλλη εβδομάδα, στις 9 Σεπτεμβρίου, για το αλκοόλ και τις εγγύους. Ελπίζω όλοι να ε, συναντηθούμε εκεί. Σας ε, καλωσορίζουμε ήδη σε αυτήν τη διάσκεψη που οργανώνουμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Ένα άλλο θέμα είναι τα ναρκωτικά. Άλλο σημαντικό τομέα. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να εγκριθούν ε, οι συστάσει του Συμβουλίου για τα προληπτικά μέτρα ή τη μείωση τη ε, κατάχρηση των ναρκωτικών από τους νέου. Και όπως γνωρίζετε, σε αυτόν τον τομέα των ναρκωτικών ε, κάνουμε ε, ε, διαβήματα για να περιοριστεί η κατάχρηση, ασχολούμαστε με την προσφορά και με την διεθνή συνεργασία. Κάπνισμα το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία, τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη. Γίνονται κινήσεις και σε εθνικό επίπεδο και σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απαραίτητο αυτό για να μειώσουμε, να μειωθεί το κάπνισμα και οι βλαβερές του συνέπειες. Ε, θα εξεταστεί η ε, πρόταση για τα περιβάλλοντα ε, χωρίς καπνό που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο και ελπίζουμε το Συμβούλιο θα μπορέσει να εγκρίνει αυτήν την σύσταση το Δεκέμβριο και υπάρχει, μπορείτε να τη διαβουλευτείτε ήδη. Ε, σας έχουμε στείλει αυτή τη σύσταση. Τώρα, ε, μια υγιής και αξιοπρεπής γύρανση. Αυτό αποτελεί μεγάλη ε, πρόκληση για μας ε, λόγω της γύρανσης του πληθυσμού και θεωρούμε ότι όλοι αξίζουν μια υγιή και αξιοπρεπή γύρανση. Ε, οι δράσεις μας σε αυτό το τομέα θα εξεταστούν από τους Υπουργούς Κοινωνικών Υποθέσεων και πρόκειται να εγκριθούν συμπεράσματα το φθινόπωρο. Αξιότιμοι βουλευτές, αγαπητέ Πρόεδρε, υπάρχουν ε, πάρα πάρα πολλά άλλα ζητήματα που θα μπορούσα να σχολιάσω, στα οποία θα μπορούσαμε να αφιερωθούμε, αλλά δυστυχώς θα πρέπει να το, τα αφήσουμε για το επόμενο τρίο Προεδριών γιατί δεν έχουμε πάρει χρόνο. Τώρα θα θέλαμε να ακούσουμε τις ερωτήσεις σας και τα σχόλιά σας και ελπίζουμε να γίνει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ τους ε, υπουργούς. Ε, πράγματι θεωρώ και εγώ πως η υγεία είναι ένα ζήτημα που απασχολεί όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως. Ε, βέβαια γι' αυτό και παρακολουθείτε με μεγάλη προσοχή από τη δική μας Επιτροπή. Έχουμε χοντρικά 40 λεπτά για να γίνουν κάποιες ερωτήσεις, για να συζητήσουμε. Αλλά επειδή θέλω να πάρουν όλοι το λόγο και έχουν ζητήσει πολύ το λόγο και οι συντονιστές, 1,5 λεπτό. Και θα πρέπει να αρχίσουν να χρησιμοποιούν αυτό το σφυράκι γιατί πραγματικά όλοι θα πρέπει να έχουν δυνατότητα να πάρουν το λόγο. Πέτερ Λίζε καταρχήν. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου και κυρία Πρόεδρε του Συμβουλίου, κάποιε πρώτε παρατηρήσει να κάνω από την δική μου πλευρά. Ε, πράγματι, η σημασία του τομέα τη υγεία αυξάνεται όλο ένα και περισσότερο και το διαπιστώνω αυτό όλα αυτά τα χρόνια που εργάζομαι σε αυτή την Επιτροπή. Ε, να πω δύο-τρία πράγματα στον κύριο Χάγκλουντ. Ε, σε ό,τι αφορά καταρχήν τα δικαιώματα των ασθενών, ε, χαίρομαι για το γεγονό ότι αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα με προτεραιότητα και ρίξτε μια ακόμα ματιά στην τροπολογία στις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί στο κείμενο του Συμβουλίου λείπουν κάποιες αναφορές που γίνονται ειδικότερα σε κάποιες πάνες ασθένειες. Επίσης, κάποιες αναφορές ηθικά ζητήματα που δεν περιέχονταν στο δικό σας ε, κείμενο και επίσης το ζήτημα των voucher, δηλαδή να μην έχουν να αντιμετωπίζουν άλλα ε, οικονομικά προβλήματα οι ασθενείς όταν ήδη έχουν λάβει την έγκριση. Σε ό,τι αφορά τώρα το φαρμακολογικό πακέτο, αυτό είναι ένα αμφιλογόμενο ζήτημα και εδώ στη δική μας Επιτροπή ε, και σίγουρα θα πρέπει να ασχοληθείτε με αυτό το ζήτημα αντιλαμβάνομαι ότι θα μπορούσε, ότι δεν μπορεί απλά να πει ε, ε, το Συμβούλιο ότι να λάβει μια θέση απέναντι στην Επιτροπή αλλά ε, θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση σε κάθε περίπτωση και σε ό,τι αφορά το, ε, την δωρεά οργάνω θα ήθελα να δώσετε προσοχή στα άρθρα 13, 14 και 15 δηλαδή σε ό,τι αφορά την άρση των περιορισμών σε ό,τι αφορά την, ε, τη δωρεά έχει γίνει μια υποχώρηση από την πλευρά της Επιτροπής οπότε θα θέλαμε να συμφωνήσετε με αυτή την υποχώρηση της Επιτροπής και ένα ακόμα ζήτημα θα ήθελα να θέσω σε σχέση με τα όσα ανέφερε ο κ. Λάνσος σε ό,τι αφορά την γρήπη δεν θα πρέπει ούτε να πανικοβληθούμε αλλά ούτε και να μην επιδείξουμε τη δέουσα προσοχή ειδικότερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στα παιδιά και συστάσεις σε ό,τι αφορά και τον εμβολιασμό και τη θεραπεία. Δηλαδή να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες ε, των παιδιών. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Ε, Δάγμα Ροτ Μπέρεν. λίγο ε, θα τα, ε, θα, πολύ σύντομα. Ε, Δυστυχώ δεν ήταν πολύ καλέ παρουσιάσει. Σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των ασθενών, δεν αντιληφθήκατε τα προβλήματα που μα αναφέρατε. Ε, είπατε ε, πεδίο εφαρμογή και στου ε, ιδιωτικού παρόχου υπηρεσιών υγεία. Είναι απλά τα πράγματα. Εάν είναι δυνατή η παροχή μια υπηρεσία υγεία σε ένα κράτο μέλο, θα πρέπει να είναι δυνατή και στο άλλο. Δεν, ξέρουμε, δεν μα ενδιαφέρει ποιο θα παράσει αυτή την υπηρεσία. Το ίδιο ισχύει σε ό,τι αφορά το ίδιο επίπεδο ποιότητα των υπηρεσιών και ασφάλεια. Εάν δηλαδή εξετάζουμε αυτό το ζήτημα διασυνοριακά, να δείτε ε, πραγματικά πόσο τρομακτικέ οι διαφορέ υπάρχουν ανάμεσα στα διάφορα κράτη-μέλη. Μην ε, θέτετε υπερβολικέ απαιτήσει. Δηλαδή, πραγματικά ε, εστιάστε στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι ίδιοι οι ασθενεί. Ε, κάποια σχόλια που έχουν γίνει από την πλευρά του Κοινοβουλίου είναι αυτό που έθεσε ο κύριο Πέτερ δηλαδή σπάνιε ασθένειε, για τι οποίε, για παράδειγμα, σε κάποια κράτη-μέλη δεν υπάρχει δυνατότητα θεραπεία. Τώρα, θα ήταν πραγματικά σκάνδαλο και θα ήταν ε, ντροπή ε, ε, το να μην αναλάβει το επόμενο ζήτημα το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά δηλαδή το φαρμακολογικό πακέτο. Για διαχωριστική γραμμή μεταξύ διαφήμισης και ε, ενημέρωση σύμφωνη. Υπάρχουν κάποια ζητήματα εδώ, αλλά υπάρχει ανάγκη ενημέρωση των ασθενών. Έχουν το δικαίωμα. Δηλαδή τα όσα αναφέρονται μέχρι στιγμή στη συσκευασία ε, δεν επαρκούν. Μένει μόνο του ασθενή. Θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό το ζήτημα και οι οργανώσει των ασθενών, εάν δεν επιληθείτε εσεί αυτού του ζητήματο, θα το πράξουν αντί για εσά. θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια συνεργασία εδώ και με αυτέ τι οργανώσει από την πλευρά των κρατών μελών και εμεί θα συνεχίσουμε τι διαβουλεύσει από την πλευρά του Κοινοβουλίου για αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ, Ντάγμα. Αντώνια Παρβάνοβα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τους δύο υπουργούς. Διαπιστώνουμε ότι είναι φιλόδοξο το πρόγραμμά σας και αυτό μας χαροποιεί διότι για αυτή την ε, θητεία θα έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε σε αυτή την Επιτροπή όσον αφορά τα θέματα δημόσιας υγείας, κάτι το οποίο δεν ίσχυσε για την προηγούμενη θητεία. Οπότε θα ασχοληθούμε με θέματα δημόσιας υγείας τώρα περισσότερο παρά ποτέ. Τα θέματα των δικαιωμάτων των ασθενών. Όπου τα είπε και η κυρία Ντάγμαρ ε, Ροτμπέρεντ, εκτός τα διασυνοριακά, είναι θέματα ασφάλειας της ιατρικών υπηρεσιών, γενικότερης ε, προσβασιμότητας, και κατά πόσο τα πιο προχωρημένα φάρμακα μπορεί κανείς να τα αγοράσει. Ένα σωρό ζητήματα τα οποία ενσωματώνονται στο χάρτη των δικαιωμάτων του ασθενείου αλλού είναι κατοχυρωμένα, σε άλλες χώρες αυτά δεν κατοχυρώνονται. Επίσης μας αναφέρατε θέματα πρόληψης και εκκρεμεί κάποια έκθεση που θα ολοκληρωθεί τέλη του έτους όσον αφορά ισότητα και υγεία θα το προωθήσετε το θέμα σε συνεργασία με την Κομισιόν λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση για να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον για, αυτή την, ε, για τις ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Επίσης, το φαρμακευτικό πακέτο είναι πολύ λεπτό το θέμα. Νομίζω ότι πασχέση με το να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των διαφόρων ε, ε, συμφερόντων, αλλά και προκειμένου είναι θέμα δημοσίου συμφέροντος. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, διακόπτει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το κύριο Σέκαρτ. Εδώ, εδώ πέρα, εδώ πέρα είμαι. Ευχαριστώ για τη σαφή σα εισήγηση, κύριε Υπουργέ. Τώρα κάτι για τα θέματα τραδία συνοριακά, γιατί βεβαίω έγινε εδώ πέρα εκτεταμένη συζήτηση, ε, ιδίω σε σχέση με το τι, τι, τι, τι, τι προποτίθεται από πλευρά εγκρίσεων. Ε, οπότε ε, εδώ πέρα θέλουμε να υπάρχει ευελιξία, ε, έχουμε επικοδομητικές ενέργειες θα πρέπει να γίνει τέτοιου είδου. Ε, να αναλυθεί τέτοιου είδου ενέργεια, ούτω ώστε να συμφωνήσει και το Συμβούλιο, να δούμε πώ θα έχουμε ευέλικτε προϋποθέσεις για να κάθε φορά να ενεργοποιείται αυτή η, ε, η, προηγουμένη έγκριση. Κυρία Γιανακουδάκη. Όχι, όχι, έγινε κάποιο λάθος, λέει η κυρία Γιανακουδάκη. Μπάσπαχ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Έχω προς και τους δύο υπουργούς, Χέγκλουντ και Λόσον, ε, κάποιες ερωτήσεις. Κύριε Χέγκλουντ πρώτα, όσον αφορά τους κανονισμούς που διέπουν τους ασθενείς, ξέρετε πάρα πολλοί συμπατριώτες μου Δανείοι πηγαίνουν στη Σουηδία, ιδίως όσον αφορά ε, τις οδοντιατρικές ε, υπηρεσίες, αλλά και πολλοί καρκινοπαθείς πηγαίνουν εκεί σας ερωτώ, αυτοί οι ασθενείς επιβάρυναν ε, το, το σύστημά σας όσον αφορά το πόσο πρέπει να περιμένει ένας Σουηδός ασθενής για τις υπηρεσίες. Επίσης, κάτι άλλο. Ε, αυτό, ε, πόσες παραπάνω ώρες εργασίας πρόσθεσε στο σύστημα. Πόσο επηρέασε. Γιατί θέλω να πω ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα επιβαρυνθεί το σύστημα παντού στην Ευρωπαϊκή να έχουμε μετακινήσεις. Κύριε Λάρσον, τώρα όσον αφορά τους ε, ηλικιωμένους. Ε, έχουμε κάποιες δραστηριότητε ή έστω και αθλητικές για του ηλικιωμένου. Γιατί ξέρετε αυτό ισχύει σε κάποιε ευρωπαϊκέ χώρε. Έχουμε κάποια συγκριτικά στοιχεία για το πώ πόσο έχει προκύψει κάποια πρόοδος, κάποιο όφελος. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος, και είναι το λόγο στην Φρανσός Γκοστέτ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ Ελληνικών Υποθέσεων, οφείλω να σας πω ότι δεν πίστηκα καθόλου σε σχέση με την οδηγία των δικαιωμάτων όσον αφορά τους διασυνοριακούς. Εγώ, ξέρετε, ε, διαδέχτηκα τον Τζον Μπάουις ε, ως εισηγήτρια και ανησυχώ γιατί δεν βλέπω να θέλετε να ταράξετε τα νερά. Μην χάνουμε το χρόνο μας. Όμως, σας πενθυμίζω με δύο λόγια ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί ότι, ότι θα πρέπει να υπάρξει ανταπόκριση σε αυτό το οποίο είπε το δικαστήριο. Έτσι απλά, τίποτα παραπάνω. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Δεν θέλουμε δυσμενεί διακρίσεις από πλευρά υγεία μεταξύ Ευρωπαίων. Αυτό που θέλουμε είναι να μπορέσει να ωφεληθεί όσο γίνεται περισσότερο ο ασθενή, για την δυνατή αγωγή ή θεραπεία. Γιατί μιλάμε για κάποιου οι οποίοι υποφέρουν. Οπότε αυτό το οποίο προσδοκώ από εσά είναι να ξεκαθαρίσετε τα θέματα του χρόνου διαγράμματο. Γιατί ε, εμείς ε, πώς και πώς περιμένουμε τι θα πείτε για την παραπίση των φαρμάκων. Βεβαίως και θα πρέπει να τα πούμε, να συνοηθούμε. Μην χάνετε χρόνο, πρόκειται για εγκληματική δραστηριότητα και εδώ θα πρέπει να, να σημειωθεί κάποια πρόοδο. Άρα χρειάζεται και εδώ πέρα αυθεντική πολιτική βούληση τώρα όσον αφορά την ε, κυρία Υπουργό. Σας υπενθυμίζω ότι στις 22 Εβδόμου εγκρίθηκε η προτάση μας ε, δύο ώστε να βοηθήσουμε την κατάσταση, την περίπτωση των, των, των ε, νόσων του, του Alzheimer, γιατί έχουμε 7 εκατομμύρια ε, ασθενείς που πάσχουν από Alzheimer στην Ευρώπη. Πρόκειται σε 20 χρόνια να έχουμε δύο φορές παραπάνω ασθενείς, επομένως θα πρέπει να φυσικά από τα κέρδα για το ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερο συντονισμό όσον αφορά την έρευνα. Παντού. Οπότε θέλω να μου πείτε, προτίθεστε και εδώ κάτι να κάνετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω δύο υπουργούς εδώ πέρα, κυρίως τον κύριο Χέγκλουμ, γιατί είμαστε και συντοπίτες. Ε, θα ήθελα και εγώ να σχολιάσω το ίδιο ζήτημα με την ε, προλαλή σα. Ε, για την οδηγία για τα δικαιώματα των ασθενών και τη διασυνοριακή περίθελψη δεν φαίνεται να υπάρχουν μεγάλες φιλοδοξίες. Το πλέον αφιλεγόμενο θέμα είναι πώς θα μοιραστεί η ευθύνη ανάμεσα στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι θα γίνει με την πρώτερη κοινοποίηση. Ε, υπάρχει ομοθυμία στο Κοινοβούλιο για αυτό το, το θέμα ε, και φυσικά και εμείς επιθυμούμε σύντομα να καταλήξουμε σε συμφωνία. Εσείς τι σκοπεύετε να κάνετε από πλευρά Συμβουλίου. Τώρα κάτι άλλο που είπε η Μαρία Λάρσον, το ακούσαμε και χτες, συγκεκριμένα πρόκειται για τον συντονισμό της δράσης, για τα εμβόλια και για την ενημέρωση για τη γρήπη. Λειτουργεί αισίως το σύστημα. Το, η Ευρωπαϊκή αυτή αρχή, η CDC και ο κύριος Γιάκοψε μας είπε διαφορετικά ε, πράγματα από αυτά που ακούσαμε στη διάσκεψη τύπου για τον εμβολιασμό. Ακούσαμε ότι ο εμβολιασμός ε, των ομάδων ε, κινδύνου θα γίνει μετά την έναρξη του εμβολιασμού των υγιών ατόμων που αρχίζει τον Οκτώβρη και πολύ μετά θα γίνει ο εμβολιασμός των ευπαθών ομάδων για να διαπιστωθεί αν δεν υπάρχουν κίνδυνοι με το εμβόλιο. Εσείς πώς το σχολιάζετε αυτό. Πώς γίνεται σε εθνικό επίπεδο να ε, διαδίδονται προφορές εντελώς διαφορετικές από αυτές που κοινοποιεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο, Ευρωπαϊκή Αρχή για τις ασθένειες αυτές. Ευχαριστούμε. Ο Κρίστοφ Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τους Υπουργούς. Θα ήθελα να επανέλθω στο ζήτημα της ενημέρωσης των πληροφοριών του κοινού για τα φάρμακα. Ε, συζητήσαμε χθες το θέμα με τον Επίτροπο Φερχόγγεν και συγκεκριμένα είπαμε ότι δεν υπάρχει βούληση από πλευράς του Συμβουλίου ούτε και ικανότητα να προαχθεί το θέμα. Ε, νομίζω ότι αυτό αξίζει να το σημειώσουμε. Ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν προτεραιότητες και θέλετε να καταλήξουμε σε συμφωνία, αλλά... Ε, δεν πρέπει να δίνετε την εντύπωση ότι θέλετε να θάψετε το θέμα. Λυπάμαι που δεν αναμένεται καμία πρόοδος στο θέμα αυτό. Ε, υποσουηδικής ε, Προεδρία. Ε, υπάρχουν ενστάσει στο Συμβούλιο, αλλά πώς να έχουμε εμείς από πλευρά Κοινοβουλίου επικοδομητική συνεργασία και να προάγουμε το ζήτημα, αν δεν γνωρίζουμε καν ε, ποιε είναι οι λεπτομερεί θέσει του Συμβουλίου, παραδείγματο χάρη για το θέμα τη διαχωριστικής γραμμή ανάμεσα στις διαφημίσεις και τις πληροφορίε. Δεν μπορεί να μην γίνεται σοβαρή ενημέρωση για όλα τα ζητήματα και πρέπει να υπάρχει σοβαρή πρόσβαση σε αξιόπιστε πληροφορίε για το κοινό. Δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε με το θέμα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι απλώς παγώνει το θέμα το Συμβούλιο. Τώρα για αυτό που είπε η κυρία Λάρσον για το κάπνισμα, θα ήθελα να ε, σχολιάζει περαιτέρω το θέμα του καπνού του Σνίσε που τον μασάμε. Äh, ε, θα ήθελα να σαν βρίσκεται εδώ μαζί μας στην ε, Επιτροπή Περιβάλλοντος και ο λόγος τώρα Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε λέει κύριε Γκούλμα και τους δύο υπουργούς για τα όσα είπαν και τα όσα απέντησαν. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία επισήμαναν θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Εγώ θέλω τώρα να σταθώ στην ασθένεια του Αλτσχάιμερ. άρα θέλω κάτι να ρωτήσω την Μαρία Λάρσεν για αυτές τις νευρο ε, ε, αυτές τις ασθένειες τέλος νευρολογικές γιατί είναι κάτι το οποίο πλήσει πάρα πολύ οικογένειες ασθενών, ασθενείς νευροεκφυλιστικές είναι αυτές οι ασθένειες 30 ε, δις ευρώ είναι το κόστος, πάρα πολλά χρήματα και εγκρίθηκαν κάποιες προτάσεις όπως ξέρετε τον Ιούλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκεί και ε, λέμε για κάποια, για κάποια έρευνα, για κάποιες επενδύσεις, για κάποια κοινή δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε, ε, επήγει το θέμα. Πέστε μας, πώς θα εξασφαλίσετε το να πετύχουμε πρόοδο σε αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Εμείς ευχαριστούμε και ο Πρόεδρος. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Καλύφθηκα από κάποιες ερωτήσεις μου από συναδέλφους και εγώ θέλω να ζητήσω διευκρινήσεις όσον αφορά την ασθένεια του Αλτσχάιμερ. Βέβαια τώρα έχουμε τις προτεραιότητες της Προεδρίας και όμως ε, είναι κάτι παραπάνω από προτεραιότητα το ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με την ασθένεια Αλτσχάιμερ. Τώρα για αυτά που είπε ο κύριος Χέγκλεντ. Πρόσεξα αυτό το οποίο σχετίζεται με την πρόσφατη δική μας δουλειά όσον αφορά τους δωρητές οργάνων είναι καλός μαθητής, αν και ο καλύτερος στην Ισπανία και οπότε με την ε, Ισπανική Προεδρία θα ασχοληθούμε περαιτέρω με το θέμα. Για τις σπάνιες ασθένειες τώρα. Πέστε μας κάτι. Με την κυρία Γκροστέτ ε, έχουμε ασχοληθεί πρόσφατα. Αλλά ε, συνεργαστής μας ήταν και ο κύριος Τρακατέλης που δεν παρίσταται πια σε αυτό το κοινοβούλιο, βουλευτής. Είναι 36, τι λέμε σπάνια, 36 εκατομμύρια είναι όλοι οι Ευρωπαίοι που πάσχουν από αυτέ τι σπάνιε ασθένειες. Επομένως, χρειάζεται καλύτερο συντονισμό. Και από πλευράς ε, των νοσοκόμων, των γιατρών, των ερευνητών. Και γι' αυτό θέλω να μου πείτε τι θα κάνετε, πώς θα δουλέψετε με κάποια συνέπεια. Γιατί πρόκειται για κάτι το οποίο πιέζει, επιτακτική προτεραιότητα. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρος. Κύριε Μισελεβάζη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργοί, εγώ τώρα θέλω να επανέλθω όσον αφορά το φρονογευτικό πακέτο στους δύο άξονες, όσον αφορά τις, την πληροφόρηση ε, στο πακέτο και προς τον ασθενή. Για να δούμε. Ας πούμε για, γιατί την για, την, ε, τι ξέρουμε, ακόμα δεν ξέρουμε τι γίνεται. Πώς θα υποχρεώσουμε τα εργαστήρια να αναφέρουν ως πληροφορίες. Δεν, δεν είναι επικοινωνία, αυτό είναι πληροφορία, πληροφόρηση. Πρέπει να δούμε ποιε είναι οι παρενέργειε, γιατί να ξέρουμε ας πούμε, το, αλουμίνιο, τη σχέση με τον Αλσχάιμερ, τι γίνεται με, το, με, με τον ε, ε, ε κλπ. Ρωτήσαμε, δεν πήραμε απάντηση. Επίση για την ενημέρωση είναι περίεργο το ότι βλέπουμε ότι έχουμε δύο μέτρα για δύο σταθμά, γιατί λέμε θα πάμε να κάνουμε μαζικό εμβολιασμό και από τη μια μεριά λέμε ότι έχουμε τι τις ομάδες πιο ευαίσθητες, τους μικρούς, τους γέρους κλπ. Και χθες όμως μίλησαμε ε, με την Υπουργό και μας είπε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτή τη σειρά γιατί δεν γνωρίζουμε αρκετά όσον αφορά τα, τα, κλινικά συμπτώματα ή τις παρενέργειες. Και τώρα ε, λέμε τέλος Νοεμβρίου. Άρα δεν υπάρχει ακόμα ε, καμία αντικειμενική ενημέρωση. Επίσης, όσον αφορά την ευθύνη, την υπευθυνότητα, θέλω να μου πείτε στη Σουηδία ποιος είναι ο υπεύθυνο για τις παρενέργειες, τα εργαστηρία, τα φαρμακευτικά. Και στη ΣΥΠΑ και αλλού δεν, δεν αρνούνται την ευθύνη των παρενεργειών των δευτερογενών επιπτώσεων ε, τα εργαστήρια. Μπά και ευθύνη είναι ευθύνη τη κυβέρνηση Τι είσαι στην Σουηδία. Η Μυροσλάβ ε, Μικολόσιτς. Μικολόσιτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ. Θα είναι πάρα πολύ σύντομος. Θα ήθελα να συγχαρώ την συνάδελφο Ριβαζίου. Διότι με κάλυψε 100% ακριβώς ήθελα και εγώ να πω τα ίδια πράγματα. Για την γρήπη ήταν έναν ή ένα. Και επίσης θέλω να ρωτήσω, ποιος φέρει την ευθύνη. Ακριβώς πάρα πολύ καλά τα είπε, γιατί τώρα μιλώ για το ποιος είναι, οι εταιρείε, ή το κράτος. Μπά και η Προεδρία μπορεί να μας ε, φωτίσει. Επίσης θα δούμε τι θα γίνει και με την οδηγία που αφορά τη, τους δωρητές οργάνων. Είμαι γιατρός και ξέρω πολύ καλά το ότι θα πρέπει να σημειωθεί κάποια πρόοδος ούτως ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτούς οι οποίοι χρειάζονται κάποια μεταμόσχευση. Που εκτιμούν πάρα πολύ το ότι η Σουηδική Προεδρία θα ασχοληθεί με τα φάρμακα. Ιδίως στις νέες χώρες μέλη. Μας καίει εμάς το θέμα στην Ανατολική Ευρώπη. Για τα ναρκωτικά. Τα ναρκωτικά είναι το θέμα μας. Ότι καταστρέφει τη ζωή πολλών νέων. Γι' αυτό και εμείς περιμένουμε κάτι, κάτι, να, να προκύψει από την Προεδρία για αυτό το θέμα. Επόμενο. Σας ευχαριστώ. Θέλω να μας πείτε λίγο κύριος Πέτρελε, το, το, το, πώς βλέπετε το ότι προσπαθούμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προσημειωθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά τη, την καταπολέμηση του καρκίνου και βέβαια είναι θέμα έρευνας, είναι θέμα του ήδη τι έχει ανακαλυφθεί και πρόσφατα λέγαμε ότι αυξάνεται η η αλληλεπίδραση της υπηρετήτας Β με τον καρκίνο του ύπαντος Θα πρέπει επομένω να περιληφθεί και αυτός ο καρκίνος στη σχετική οδηγία που θέλετε να αναθεωρήσετε. Κατάχρηση του αλκοόλ, ε, και αυτό βέβαια είναι ένα φαινόμενο το οποίο ε, σχετίζεται με αυτόν τον καρκίνο. Άρα θέλω να τι πιστεύετε και για αυτά τα θέματα. Κυρία Εστρέλα, ευχαριστώ. Θα ήθελα να σχολιάσω την ε, οδηγία για την παροχή διασυνοριακής περίθελψης. Θέλω να τονίσω συγκεκριμένα την ε, σημασία της πρώτερης έγκρισης, πρώτερης άδειας. Όχι μόνο για να κατοχυρωθεί η ασφάλεια για τον ασθενή, αλλά ταυτόχρονα για να κατοχυρωθεί η βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας των ε, κρατών μελών όπου υπάρχουν εθνικές υπηρεσίες υγείας δωρεάν και καθολικές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το τόνισε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη σχετική εκθεσή του. Κάτι άλλο τώρα που σχετίζεται με τα εμβόλια. Ε, αναφέρθηκε ήδη το ζήτημα από τους συναδέλφους. Απλά ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας ε, στα διάφορα δημοσιεύματα που δεν έχουν διαψευστεί, που λένε ότι ενδέχεται να υπάρξουν πάρα πολλοί βλαβερές παρενέργειες ε, από τα εμβόλια ακόμη και για τους υγιείς ανθρώπους και αναρωτιούνται οι πολίτες ε, μήπως είναι πιο επικίνδυνο το εμβόλιο από την ίδια τη γρήπη. Μη, το Συμβούλιο μπορεί να δώσει εχέγγυα για την ε, ποιότητα και για την ασφάλεια των εμβολίων, διότι από ό,τι λέγεται δεν υπήρξε χρόνος για να γίνουν οι απαιτούμενες δοκιμές. Τέλος, κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ τη Σοηδική Προεδρία για την, το βάρος που θα ρίξει στο θέμα της κατάχρησης ε, του αλκοόλ ε, κυρίως από τους νέους. Ε, συγχαρητήρια για την διοργάνωση της διάσκεψης και αναμένουμε με ανυπομονησία τα αποτελέσματα αυτών των εργασιών. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη διότι μισό Ριβαζή ως επιτοπλίστων με κάλυψε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και ζηγίζω αυτά τα οποία σας λέω Όταν Θεωρούμε ότι είναι δυνατόν να μην υπάρχει πανευρωπαϊκή ενημέρωση όσον αφορά το εμβόλιο για, το, για την γρήπη τα έναν ή ένα. Μα τι αξιοπιστία έχουν οι εθνικέ αρχέ, τι θα είχαν ω αξιοπιστία, εάν βρισκόντουσαν σε κατάσταση αντίφαση μεταξύ του, εάν δεν είχαν κάποιο είδου έγκριση με το ε, με το ECDC και επομένως αυτό θα ισχύει και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευρά πληροφόρηση. Είδατε τι είπε η κυρία εδώ όσον αφορά το, το, τον κίνδυνο, όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού. Κάτι το οποίο είναι μείζον πάρα πολύ σημαντική κοινωτική πολιτική. θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση του κόσμου για τα θέματα της υγείας. Αν λοιπόν δεν έχουν τέτοια πολιτική, τι να πούμε για τις άλλες πολιτικές. Μουτιέρες Κορτίνς, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Με δύο λόγια θα σας πω τα εξή. Τα δύο θέματα που με απασχολούν. Κινητικότητα των ασθενών. Εγώ ε, συμφωνώ, συμφωνώ, στηρίζω με την νομοθεσία και συμφωνώ με αυτό που προσβεύει το Κοινοβούλιο και όχι το Συμβούλιο. Είναι σκάνδαλο αυτά που λέει το Συμβούλιο για τις προτάσεις της Κομισιόν. Είπαμε ότι ε, θέλουμε να, το θέμα να διεκπαιρεωθεί, ε, ξέρουμε ποιες είναι οι ενστάσεις ισπανικές, ε, άρα θα πρέπει να, κάτι να κάνει η Σουηδική Προεδρία γιατί μετά η Ισπανική θα το κλείσει το θέμα, θα το, θα, θα το, δεν θα το διεκπαιρεώσει. Άρα, αυτό θα πρέπει να δούμε που είναι θέμα κλειδί. Οι δεπάνες δε ιατρικές. Περιπτωσιολογικά κρίνεται το θέμα του κόστους. Και θα πρέπει να αποφασίζει αυτός ο οποίος πληρώνει. Έχω δύο συγγενείς μου μέσα στην οικογένεια που πάθανε αυτή την γρήπη. Το λέμε ήταν μικρό κοριτσάκι και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο συμβαίνει και δεν είναι η γρήπη προ το παρόν, δεν είναι κάτι τόσο βαρύ. Το θέμα είναι ε, η διάγνωση. Γιατί στην Ισπανία και στην περισσότερη Ευρώπη τα κέντρα υγεία δεν έχουν τις ε, αναγκαίες ουσίε τα αναγκαία σκευάσματα για την διάγνωση. Επομένω πρέπει κανεί να φτάσει σε προχωρημένη κατάσταση ασθένεια για να το διαγνώσουν. Βέβαια, αυτή η ελαφρία γρήπη μπορεί να γίνει πνευμονία. Άρα να κάτσουμε και σοβαρά να δούμε όλη αυτή τη διαδικασία, ακόμα και τη διάγνωση που είναι πάρα πολύ σημαντικό και ακόμη πιο σημαντικό μια που δεν φύγεται το θέμα αρκετά. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε ένα εύρυθμα λειτουργών σύστημα υγείας ε, προϋποθέτει ότι οι δαπάνε οι οποίες ε, προκύπτουν από τη διασυνοριακή περίθαλψη ασθενών ε, πράγματι αναλαμβάνονται από τα εκάστοτε κράτη-μέλη. Και ακριβώς το πρόβλημα για το για κάποια κράτη-μέλη που έχουν ένα καλό τέτοιο σύστημα είναι να δημιουργούνται τέτοιε υψηλέ δαπάνε. Οπότε να ε, καταστεί δυνατό μέσω ενός συστήματος ε, του να καταβάλλονται δαπάνες από τα αρμόδια κράτη-μέλη στα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία υποδέχονται ασθενείς. Σε ό,τι αφορά ε, εκείνο τώρα το σύστημα της εκ των προτέρων έγκρισης, της προέγκρισης, έχετε σκεφτεί κάποιους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε αυτό να καταστεί το σύστημα δηλαδή λίγο πιο αποτελεσματικό χωρίς να είναι απαραίτητη η, καταβολή υψηλών ταπανών. και μετά, σε ό,τι αφορά το αλκοόλ, έχει πραγματικό νόημα η διοργάνωση μιας διάσκεψη για αυτό το ζήτημα. Εγώ αναφέρω ε, ενδεχομένως ε, και το ζήτημα των νέων, ε, δηλαδή το πρόβλημα του αλκοόλ που αφορά όλο και περισσότερο τους ε, νέου. Μήπως θα μπορούσε πέρα από τα όσα πράττει ήδη να κάνει κάτι παραπάνω, κάτι πιο ουσιαστικό η Συνδική Προεδρία σε σχέση με το αλκοόλ. Θα πω δύο λόγια σε σχέση πάλι με την γρήπη τα κάτω τον όσων είπαν η συναδελφή θα μας απασχολήσει έτσι καλώς και τα επόμενα χρόνια και έχουμε τη Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας και πριν από λίγες μέρες έσωθε το ερώτημα τι χρειάζεται περισσότερο όσον αφορά την καταπολέμηση αυτή της γρήπης. Τη ρωτήσανε και αυτή τι είπε, τι, τι απάντησε. Χρειάζεται πολιτική ηγεσία. Χρειάζεται η πολιτική ηγεσία να βρει το σωστό συντονισμό και νομίζω ότι εσείς ε, από τη θέση που θα έχετε τους αμέσως επόμενους μήνες θα πρέπει να ε, αντιμετωπίσετε ως αναγκαιότητα αυτό το, το ρόλο, τον πρωτοπόρο που έχετε αναλάβει για κάποια εκκρεμή ιατρικά ζητήματα. Γιατί ακόμα εκκρεμούν πάρα πολλά ερωτηματικά, όπως ας πούμε αυτό για, για τις δευτερογενείς συνέπειες, για τις ε, αντενδείξεις, για, για τις ε, όλες τις συνέπειες του, εμβολιασμού, όπως ακριβώς το είπε και αυτή η διευθύντρια του ΠΟΕ, του, συγγνώμη, του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας. Να 150 εκατομμύρια εμβόλια για 6 δις, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο ε, ανθρώπους. Όταν ξέρουμε αυτό μας τα λένε και οι ειδικοί, γιατί πρόκειται για ένα σωρό ε, κόσμο που ποιος αν πάθει πνευμονία, το 40% αυτούς θα πεθάνει. Επομένως, εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα ερωτήματα, αφορούν την ενημέρωση και απαιτούν απαντήσεις. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, τα ζητήματα που αφορούν την πανδημία ε, συνεχίζουν να μας απασχολούν και δεν μπορούν να απαντηθούν κάποια από τα ερωτήματα που κρεμούν ακόμα, αλλά αναφερθήκατε ε, και στις δυνατότητες ε, προμήθειας εμβολίων για τα κράτη-μέλη τα οποία ακόμα δεν έχουν ζητήσει Αντίστοιχε ποσότητες από τους κατασκευαστέ. Υπάρχουν βάσιμε ανησυχίε να μην υπάρχουν επαρκή αποθέματα εμβολίων, δηλαδή να μην υπάρξει επαρκή σε παραγωγή. Τι προτίθεται να κάνει το Συμβούλιο ή η Επιτροπή ούτως ώστε να έχουμε πράγματι επαρκή ποσότητα εμβολίων και πώ ε, τα εμβόλια αυτά θα διανεμηθούν, πώ θα κατανεμηθούν στα κράτη-μέλη. Γιατί βέβαια και αυτό θα αποτελέσει κάτι το οποίο, ε, με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθείτε. Ε, κυρία Λάρσεν, έχετε ε, βέβαια ε, να αντιμετωπίσετε και την, ε, αφού αυτό σε και στις αμμοδιότητες του Υπουργείου σας την τρίτη ηλικία. τρίτη ηλικία συγγνώμη. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη σήμανση των τροφίμων θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας και ακριβώς στην, στις μεγαλύτερες ηλικίε, δηλαδή να έχουμε εδώ σαφή σήμανση, ευδιάκριτη, κατανοητή ούτω ώστε να μπορούν και οι άνθρωποι σε μεγαλύτερες ηλικίε να αγοράζουν τα τρόφιμα που θέλουν. Δηλαδή να το δούμε ως προτεραιότητα αυτέ τις μεγαλύτερες ηλικίες. Ε, σε ό,τι αφορά το αλκοόλ. Ε, να μην ε, κάνουμε εδώ λανθασμένες, λανθασμένη χρήση των εκφράσεων, να μην μιλάμε για χρήση του αλκοόλ. Κατάχρηση πάντα πρέπει να λέμε ε, σε σχέση με το αλκοόλ. Εντάξει, ε, άλλο το, το ζήτημα της κουλτούρας που υπάρχει στην ε, Ευρώπη, δηλαδή με την κατανάλωση ενός ποτηριού κρασιού μαζί με το φαγητό, αλλά άλλο πράγμα αυτό και άλλο η κατάχρηση του αλκοόλ, ειδικότερα για παράδειγμα σε δίωση σε άλλες τέτοιες ομάδες. Αυτά. Ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ζήτησα το λόγο, λόγω των όσων είπατε, σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι δεν θέλετε να συνεχίσετε με ε, το πακέτο σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των ασθενών. Σας λέω λοιπόν ότι εγώ ε, διαφωνώ κατηγορηματικά ε, και σας το λέω ανοιχτά, δηλαδή εγώ χρειάζομαι να... Είμαι, είμαι απόλυτα υπέρ ενός τέτοιου συστήματος και δεν μπορούμε να πάρουμε ένα τέτοιο σύστημα όπως το σύστημα ΦΑΣ, το οποίο έχουμε εξευρωπαίσει, ποιο τελικά θα ταχθεί υπέρ αυτού του συστήματο, αν όχι εσεί, αν όχι η Σουηδική Προεδρία. Ε, εγώ άκουσα και ε, χθεσινή επίσκεψη που είχα από την κυρία ότι είναι η Σουηδική κυβέρνηση υπέρ και σας λέω πως δεν υπάρχει ε, καμία καλύτερη ευνοϊκότερη συγκυρία από τη σημερινή εδώ και 10 χρόνια για να καταφέρουμε κάτι. Δηλαδή πήραμε κάτι από το σουηδικό επίπεδο, το εξευρωπαίσαμε και τώρα το καταργούμε, καταργούμε όλη αυτή την προσπάθεια επειδή δεν έχετε επιτύχει την πλειοψηφία που χρειάζεται στο Συμβούλιο. Συνεχίστε να προσπαθείτε, συνεχίστε να εργάζεστε προς αυτό το στόχο για να επιτύχετε πλειοψηφίε μέσω συμβιβαστικών λύσεων. Όπως κάνουμε και εμείς στο Κοινοβούλιο. Γιατί αυτό που δεν θέλουμε να γίνει είναι να μην θέλουμε τελικά το 2009, μέσα στο έτος 2009, έναν ασθενή ο οποίος είναι ενημερωμένος. Ένα Ελληνί ο οποίο είναι υπεύθυνο. Δεν είναι ζήτημα ηθικής εδώ. Είναι ένα ζήτημα των, ε, ε, α, των ταμείων των Ταμείων Δημόσια Ασφάλιση τη Υγεία, δηλαδή που λένε τι, ότι δεν επιθυμούν ένα τέτοιο ενημερωμένο, καλά ενημερωμένο ασθενή, γιατί είναι υπερβολικά ακριβώ. Αυτό λένε, ε, δεν μπορεί να γίνεται κάτι τέτοιο το 2009. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Είχαμε εδώ ένα μαραθώνιο από ερωτήσει. Πόσο εμπειρογνώμονε έχουμε εδώ στην Επιτροπή μα, πόσο μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει για τα ζητήματα. Ε, Ευχαριστώ. Πάρα πολλές ερωτήσεις. Ε, ελπίζω να βρω ε, συμβατές απαντήσεις από τον κατάλογο που έχω για να σας δώσω. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο ότι πολλούς σας απασχολεί το θέμα της διασυνοριακής περίθαλψης και των δικαιωμάτων των ασθενών. Επίσης, ε, άλλους απασχολεί το θέμα των φαρμάκων και μία τρίτη κατηγορία είναι η δωρεά οργάνων. Αυτά, αυτές είναι οι τρεις κατηγορίες ε, που ε, ενδιαφέρουν περισσότερο τους βουλευτές. Θα προσπαθήσω εν συντομία να σας δώσω κάποιες απαντήσεις. Για την κινητικότητα των ασθενών, όπως είπαν πολλοί βουλευτές και όπως είπα και εγώ στην εισαγωγική μου παρουσίαση, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα και από πλευρά της Προεδρίας ε, έχουμε αυτήν την μοναδική φιλοδοξία να προωθήσουμε το θέμα το φθινόπωρο. Δεν έχουμε άλλη τόσο σημαντική φιλοδοξία. Έχουμε ακούσει διάφορες επιχειρηματολογίες από κράτη-μέλη που έχουν πολλά και διαφορετικά προβλήματα. Ε, η δική μας δουλειά είναι να επεξεργαστούμε τα δεδομένα και να δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε ε, σε μία πρόταση την οποία θα υποβάλουμε στη δεύτερη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο. Πρέπει, χρειαζόμαστε όμως πλειοψηφία στο Συμβούλιο ε, και εμείς με την ιδιότητα του Προέδρου θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε αυτή την πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα ε, στα δικαιώματα των ασθενών ε, για διασυνοριακή περίθαψη με ασφαλή τρόπο και των εθνικών συμφερόντων, δηλαδή των συμφερόντων των κρατών ε, να κατοχυρώσουν τα συστήματα υγείας τους και κοινωνικής ασφάλισης. Πρέπει να βρεθεί αυτή η ισορροπία. Ακούσαμε διάφορα σχόλια και θα ήθελα να αρχίσω σχολιάζοντας ε, το θέμα των vouchers, των δελτίων. Ότι δεν χρειάζεται δηλαδή ο ασθενής να καταβάλει κάποιο ποσό. Μα δεν γίνεται αλλιώς. Αλλιώς ε, θα έχουμε ένα σύστημα που θα λειτουργεί μόνο για τους πλούσιους. Δεν θα λειτουργεί για αυτούς που έχουν χαμηλό εισόδημα. Είναι ζωτική σημασία σε αυτό το θέμα των δελτίων. Και φυσικά επεξεργαζόμαστε εντατικότατα ε, τη λύση για αυτό το ζήτημα. Άλλες ερωτήσεις έφεραν επί της πρώτερης έγκρισης, πρώτερης άδειας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το ζήτημα. Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά συμφέροντα στο Συμβούλιο και ο στόχος μας είναι να σταθμίσουμε τις θέσεις για να καταλήξουμε ναι μεν σε συμφωνία αλλά και ταυτόχρονα να καλύψουμε ε, τα, τα δικαιώματα των ασθενών, ε, δηλαδή να κινούνται ελεύθερα οι ασθενείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διάφοροι βουλευτές δήλωσαν απογοητευμένοι σε σχέση με το μέλλον, μα και εγώ ε, το ίδιο νιώθω, ε, θα προσπαθήσω ε, κατά τη διάρκεια της Ειδικής Προεδρίας να προωθήσω αυτά τα ζητήματα, αλλά μόνοι μας δεν πρόκειται να τα καταφέρουμε. Χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας και σας ξαναλέω, χρειάζεται πλειοψηφία, αλλιώς δεν κινείται τίποτα στο Συμβούλιο. κατόπιν. τα φάρμακα. Έχουμε στα τρία διακριτά τμήματα του πακέτου για τα φάρμακα τι να σας πω, στο Συμβούλιο δεν υπάρχει τρόπος υπό Προεδρίας να προωθήσουμε το θέμα για την ενημέρωση των ασθενών. Αποκλείεται να επιτύχουμε πλειοψηφία κατά τη διάρκεια του εξαμένου της Προεδρίας και γι' αυτό και εμείς αποφασίσαμε να εστιάσουμε την προσοχή μας στα δύο άλλα τμήματα που επίσης είναι σημαντικά. Μα και εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι είναι σημαντική η ενημέρωση των ασθενών. Υπό Σουηδικής Προεδρίας ξαναλέω δεν υπάρχει ε, πιθανότητα να ευοδοθούν οι προσπάθειές μας για αυτό και θα ασχοληθούμε με τα άλλα δύο τμήματα και εδώ τίθενται διάφορα ζητήματα διαφορετικού χαρακτήρα μεταξύ των οποίων το ότι υπάρχουν συνταγματικού χαρακτήρα προβλήματα σε διάφορα κράτη-μέλη. Ε, ξέρετε πώς λειτουργούν ε, οι δημοκρατίες. Δεν γίνεται εμείς να βρούμε λύση μέσα σε έξι μήνες. Ε, πρέπει να γίνει προσεκτική προετοιμασία εάν χρειαστεί αλλαγή του συντάγματος. Ε, πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε άλλη διέξοδο από αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, τα ζητήματα για τα σπάνια φάρμακα. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτού του τομέα. Ας αρχίσω με τις σπάνιες νόσους, λοιπόν, καλύτερα. Τα κράτη-μέλη μέσα από τις συστάσεις του Συμβουλίου για τις Σπάνιες Νόσους έχουν συμφωνήσει ότι υφίσταται ανάγκη για αυξημένο συντονισμό, αυξημένη συνεργασία. Παραδείγματο χάρη για τι βάσει δεδομένων, για να ε, ε, βρίσκονται οι γνώσει για τι σπάνιε γνώσει εύκολα. Ε, είναι πρόωρο ακόμη, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς μπορούμε να κινήσουμε το θέμα. Για τις σπάνιες νόσου. η Σουηδία έχει αναλάβει πρωτοβουλία για, την, για ένα πιλωτικό πρόγραμμα για τα φάρμακα αυτά. Ε, έγινε και διάσκεψη 29 Ιουλίου ε, στη Στοχόλμη για αυτό το θέμα και συμφωνήθηκε ότι θα αρχίσει να τρέχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα για συλλογή δεδομένων και ανταλλαγή γνώσεων σχετικά ε, με τις παρενέργειες αυτών των φαρμάκων και το φθινόπωρο θα συνεχιστεί. Θα υπάρχει συνέχεια αυτής τη διάσκεψη στα πλαίσια του πιλωτικού προγράμματος ε, και όλοι δικαιούνται τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη και αν δημιουργήσουμε ένα δίκτυο ανταλλαγής καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη θα είναι η προστιθέμενη αξία αν διασυνοριακά συνεργαστούμε για να καλύψουμε τις ανάγκες αυτών των συμπολιτών μας. ένα λεπτάκι να δω αν υπάρχουν κάποια άλλα ζητήματα που σχετίζονται με αυτό. Πολλά ακούσαμε για, τους, ε, για τα εμβόλια, αλλά η Μαρία Λάσον θα απαντήσει. Συγγνώμη. Α, μου θυμήσατε μπράβο, τα όργανα, η δωρεά των οργάνων. Λοιπόν, δωρεά οργάνων. Εδώ έχουμε στενή συνεργασία με τους Ισπανούς συναδέλφους μας. Ε, γιατί όπως ακούσαμε είναι και καλύτεροι μαθητές στον τομέα αυτό. Σχετικά με την βούληση των ε, συμπολιτών μας να γίνουν δωρητές οργάνων. Στην, ε, στην Ισπανική Προεδρία λοιπόν θα, θα σημειωθούν μεγάλες εξελίξεις σε αυτό το τομέα. Ο στόχος είναι να βρούμε έναν ασφαλή τρόπο ώστε να γίνονται οι δωρεές οργάνων και γνωρίζουμε ότι σε πολλά κράτη-μέλη πρέπει να γίνουν ε, εσωτερικά μεγάλα βήματα ούτω ώστε να υπάρχει αυτή η θέληση σε επίπεδο πολιτών να γίνουν δωρητέ οργάνων. Σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν πολλά να γίνουν ακόμη, αλλά και σίγουρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να συντονίσουμε τι δράσει μα. Αλλά ο στόχο γενικά είναι η ποιότητα, η ασφάλεια που πρέπει να διέπει την διαδικασία δωρεάς οργάνων. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείχνετε, τη δέσμευσή σας. Άκουσα μία σειρά από ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω την δυνατότητα να σας μιλήσω. Ελπίζω να είναι σαφής οι απαντήσεις μου. Θα ομαδοποιήσω αυτές τις ερωτήσεις. Πολλές φέρουν επί της γύρανσης και άλλες επί της γρήπης. Θα αρχίσω με αυτές. Αρχικά να σας πω ότι... Υπάρχει αυτή η τάση για δημογραφική γύρανση. Ε, αυτό σημειώνεται ως τάση σε όλα τα κράτη-μέλη. Μα αυτό είναι φανταστικό γιατί σημαίνει ότι υπέτυχε το κράτος πρόνοιας και πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτή την εξέλιξη. Βέβαια, ταυτόχρονα πολλοί οι ηλικιωμένοι είναι υγιείς, ενεργοί και πρέπει και εμείς να τους ε, σπρώχνουμε να ενεργοποιούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην αγορά εργασίας γιατί ξέρετε ότι προάγει και την υγεία τους το να συνεχίσουν να εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα επίσης. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ε, ούτως ώστε να παρέχουμε την κατάλληλη περίθαλψη χρειάζονται οι ηλικιωμένοι και υπάρχουν πολλοί που υποφέρουν από νευροεκφυλιστικές νόσους μεταξύ των οποίων και το Αλτσχάιμερ. Η περίθαλψη των ηλικιωμένων είναι ως επιτοπλίστων ένα εθνικό θέμα. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, αλλά εγώ είμαι πεπισμένη ότι μπορούμε να έχουμε σημαντικά κέρδη από μια συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο με σαφέστερο τρόπο σε σχέση με το παρελθόν και γι' αυτό χαίρομαι ότι, ε, για τη συνεργασία που είχαμε στην Τρόικα με, την, ε, με τις προηγούμενες προεδρίες για το θέμα των ηλικιωμένων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που ε, τίθενται αυτά τα ζητήματα και γράφονται στην ημερήσια διάταξη της Ένωσης και ο στόχος που έχω για την Προεδρία μας είναι τα θέματα των ηλικιωμένων να εγγραφούν με πιο μόνιμο τρόπο τρόπο, αν θέλετε, στην ημερήσια διάταξη της Ένωσης και γι' αυτό θεωρώ ότι χρειαζόμαστε περισσότερες συγκρίσιμες στατιστικές ε, για ε, τις παρεμβάσεις που γίνονται, παραδείγματος χάρη, για την βελτίωση της υγείας των ηλικιωμένων ε, και τα αποτελέσματα των διαφόρων δράσεων ως προς την κοινωνική πρόνοια και την υγειονομική περίθαλψη. Θα επιδιώξουμε να εγκριθούν αποτελέσματα από το Συμβούλιο το Δεκέμβριο ε, και θα έχουμε κατευθυντήριες γραμμές φυσικά από τη διάσκεψη των εμπειρογνωμών που θα γίνει το Σεπτέμβριο. Να μένω με ανυπομονησία τη συνεργασία με το Κοινοβούλιο και ξαναλέω ότι θέλουν αυτά τα ζητήματα να συζητούνται με πιο μόνιμο τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πρέπει να βρούμε ένα κοινό τρόπο για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Ε, χρειαζόμαστε συντονισμένη δράση για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η υγειονομική περίληψη των ηλικιωμένων στο μέλλον. Ας περάσω στη γρήπη τώρα. Ε, ε αυτό το ζήτημα φυσικά το παίρνουμε πάρα πολύ στα σοβαρά διότι δεν έχουμε χρόνο ε, και γι' αυτό συγκαλούμε αυτό το έκτακτο συμβούλιο με μοναδικό σημείο στη μέση διάταξη τη γρήπη. Δηλαδή, τουλάχιστον αυτό μπορούμε να προβλέψουμε μέχρι στιγμή. Γι' αυτό συγκαλέσαμε το έκτακτο συμβούλιο. Είναι ζωτική σημασία στο θέμα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε το συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Είναι κάτι που πρέπει να μα απασχολήσει ήδη τώρα. Σε αυτό το τομέα, και είναι σημαντικό να το πω, ε, υπάρχει ε, αρμοδιότητα μεγάλη των κρατών μελών. Έχουμε προετοιμαστεί με πολλούς και διάφορους τρόπους. Ε, υπάρχει η κοινή Ευρωπαϊκή έρχη για τις μεταδοτικές ασθένειες, η οποία έδωσε καλές συμβουλές σε όλα τα κράτη-μέλη για να καταρτήσουν τα εθνικά σχέδια δράσης αντιμετώπισης της γρήπης. Αλλά φυσικά μπορούμε να συνεργαστούμε περαιτέρω και είναι προφανές ότι θα προκύψει τη θέμενη αξία από την Ευρωπαϊκή Συνεργασία. Για την παγκόσμια διάσταση έχουμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Οργανισμό Υγείας ε, και πρέπει να ε, λειτουργούμε βάσει των ε, συστάσεων του ΠΟΕ, ακόμη και σε ΠΟΗ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ακόμη και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Μάργαρετ Τσάντα έχει μας μίλησε για τον ηγετικό ρόλο και φυσικά υπάρχει βούληση από πλευράς του κρατών Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προωθήσουμε κάποια ζητήματα. Απλά χρειαζόμαστε μία συγκεκριμένη στρατηγική και ελπίζουμε στις 12 Οκτωβρίου να εγκριθεί αυτή η κοινή στρατηγική. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα που πρέπει να συζητήσουμε. Τα ανέφερα στην παρουσίασή μου. Σας μίλησα για τα επικοινωνιακά θέματα. Το ανέφεραν και οι βουλευτές και χαίρομαι που στο ξενοδοχείο που είμαι εδώ στις Βρυξέλλες ε, βλέπω ότι έχει φτάσει εκεί το χέρι της ECDC και έχει βάλει μία φύσα που περιγράφω τα διάφορα μέτρα για την αντιμετώπιση της ε, γρήπης θεωρώ ότι μπορούμε και σε εθνικό επίπεδο να επιφέρουμε κάποιες βελτιώσεις ε, πέρα από την κοινοτική πολιτική. Χρειάζεται καλύτερη επικοινωνιακή πολιτική γενικά. Επίσης, σας μίλησα για την παγκόσμια αλληλεγγύη. Ε, δηλαδή, αν δεν φτάσουν τα εμβόλια, πρέπει να έχουμε μια αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Επίση, κοινή διαχείριση τη μεταπόληση των εμβολίων ανάμεσα στι χώρε. Ε, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να διαχειριστούμε αυτό το θέμα γιατί υπάρχουν ναι, δυσκολίες ε, νομικού χαρακτήρα αλλά τα ζητήματα τα οποία επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα για να υποβάλει την πρότασή της ε, μας απασχολούν και φυσικά θα συνεχίσουμε εμείς να συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τα εμβόλια, την ασφάλεια των εμβολίων και τον εμβολιασμό τώρα. Είμαι πεπισμένη ότι λειτουργούν αισίως οι διατάξεις του συστήματος ασφάλειας. Κατοχυρώνεται η ασφάλεια από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων στο Λονδίνο, αλλά υπάρχουν και άλλα επιπρόσθετα συστήματα ελέγχου. Όταν είναι έτοιμο και εγκριθεί το εμβόλιο, θεωρώ ότι μπορούμε να αισθανόμαστε ασφαλείς. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Πρέπει να ε, περιμένουμε βέβαια να δούμε και τα αποτελέσματα αυτών που θα το δοκιμάσουν το εμβόλιο και πρέπει να δούμε και τις συστάσεις που θα συνοδεύσουν το εμβόλιο για τον εμβολιασμό των παιδιών παραδείγματο χάρη. Κάτω από τα τρία έτη έχουν ήδη πει οι ειδικοί ότι πρέπει να περιμένουμε. Δεν ε, ε, θα πρέπει ακόμη να τα εμβολιάσουμε τα παιδιά και μετά μπορούμε να καταβούμε ως τους έξι μήνες για τον εμβολιασμό των παιδιών. Πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθήσουμε τις συστάσεις που θα συνοδεύσουν τα νέα εμβόλια και οι εθνικές αρχές πρέπει με ενεργό τρόπο να συνεργάζονται και με το ECDC, την Ευρωπαϊκή Αρχή για τις Μεταδοτικές Ασθένειες και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μπορεί να προκύψει διάσταση απόψεων, αλλά... Κοιτάξτε, εγώ αυτά που έμαθα ότι είπε το ECDC χτες δεν είναι αυτά που άκουσα από εσά. Δηλαδή δεν βλέπω αντίθεση ανάμεσα σε αυτά που λέει το ECDC και αυτά που λένε οι Σουηδικέ αρχέ για αυτά τα ζητήματα, ξέρετε, πάντοτε έτσι είναι, δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις. Τι να κάνουμε, πρέπει να το δεχτούμε ότι εκ των υστέρων ε, θα πάρουμε κάποιες άλλες απαντήσεις, έτσι έχουν τα πράγματα. Πάντως, ε, αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στο ζήτημα και σας είπαμε ότι θα συγκαλέσουμε έκτακτο συμβούλιο για αυτό το θέμα για να δούμε σε ποιους τομείς μπορεί η ευρωπαϊκή δράση, ο ευρωπαϊκός συντονισμός να προσφέρει τη θέμενη αξία. Και όταν υπάρχουν ε, οι δυνατότητες ε, θα γίνουν ευρύτατοι εμβολιασμοί. Για το αλκοόλ, ε, ευτυχώ που είναι σημαντικό το θέμα για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι έχουμε πολύ μεγάλα ποσοστά κατανάλωση αλκοόλ στην Ευρώπη σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο και ήταν πάρα πολύ σημαντικό Ενδιαφέρουσε οι συζητήσεις στο Συμβούλιο Υπουργών. Ε, δηλαδή υπάρχει σχετικά μεγάλη ομοθυμία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ε, το αλκοόλ είναι θέμα δημόσιας υγείας και πρέπει να το αποδώσουμε μεγάλη σημασία, κυρίως ως προς την κατάχρηση του αλκοόλ από τους νέους. Ε, και ζητούνται δραστικά μέτρα ε, και από την διάσκεψη των εμπειρογνωμόνων ε, και θα δούμε αν θα είναι τελικά ε, δυναμική η δράση που θα αναλυθεί ανάλογα με τα συμπεράσματα που θα εγκριθούν από το Συμβούλιο. Αντώνια Πανανόβα με ρώτησε κάτι για τα θέματα δημόσιας υγείας. Ε, και ότι θα αναμένεται ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ποιότητα της υγείας. Ναι, το Δεκέμβριο θα εκδοθεί η ανακοίνωση, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε εμείς να επιληφθούμε του ζητήματος υποσυδικής προεδρίας. Και τέλος, Κριστόφερ Φιέλνερ μου μίλησε για το σνίσο, ε, για αυτό τον καπνό που βάζουμε στο στόμα. Αυτό του αυτός ο καμνό δεν θα μας απασχολήσει. Λοιπόν, θα σου απαντήσω τηλεγραφικά, Κριστόφ. Δεν θα μας απασχολήσει στην Προεδρία μας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ του δύο υπουργού, ε, του δύο προέδρου ε, του Συμβουλίου. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με αυτά τα ζητήματα, καθώς πραγματικά ενδιαφέρουν πάρα πολύ την Επιτροπή μα. Ε, ε, και αναμένουμε να δούμε και τι θα γίνει από δική σας πλευρά γιατί πραγματικά αναμένουν οι πολίτε της Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι να γίνει. Ε, η συνεδρίασή μας ολοκληρώθηκε, θα ειδωθούμε ξανά στι 30 Σεπτεμβρίου. Γεια σας.